Dear colleagues. Αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω μπορούμε να ξεκινήσουμε με την ψηφοφορία. Να υπενθυμίσω στους συναδέλφους ότι θα ψηφίσουμε ηλεκτρονικά. Πρώτη ψηφοφορία για το σημείο αυτό 7. Υποχρεωτική αναγραφή χώρας καταγωγής ε, ή τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα. Άρχεται η ψηφοφορία. Ψήφισαν όλοι. Όχι. Καλά. Πρέπει να περιμένουμε ένα συνάδελφο. Όχι, ακόμα. Εντάξει, αν έχουν ψηφίσει όλοι, πέρας τη ψηφοφορία. Εγκρίνεται. Τώρα μπορούμε να περάσουμε στη δεύτερη ψηφοφορία για την επιθυμία του Ουζίκα. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε ψηφοφορία. ομόφωνη ψήφος. Okay, now we... Ωραία. Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε τη συζήτηση για το σχέδιο ψηφίσματος για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής ή του τόπου προέλευσης για ορισμένα τρόφιμα. Πρόκειται για το σημείο 9 στην ημερήσια διάταξη. Θα δώσω απευθεία το λόγο στους συνεισηγητές, η Γκλένις Βίλμοντ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Έχει περάσει ένα χρόνος από τότε που ενέκρινε το Κοινοβούλιο ψήφισμα ζητώντας υποχρεωτική επισήμανση της χώρας καταγωγής. Και Χαίρομαι που θα ξεκινήσει η εφαρμογή του στη Γαλλία. Θεωρώ ότι αποτελεί ένα βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση, αλλά είμαι απογοητευμένη διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή αρνείται να διασφαλίσει ότι όλοι οι καταναλωτές στην Ευρωπαϊκή Ένωση θα έχουν αυτές τις πληροφορίες. Με το ψήφισμα αυτό ε, ουσιαστικά δεχόμαστε κάποια από αυτά τα οποία προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ζητάμε υποχρεωτική αναγραφή για μεταποιημένο κρέας και τα γαλακτοκομικά. Ε, είναι τα προϊόντα για τα οποία οι καταναλωτές ενδιαφέρονται περισσότερο για την αναγραφή της χώρας καταγωγής και ε, δεν θα είναι λογικά και πολύ δύσκολο να παρέχονται αυτές οι πληροφορίες. Ήδη κάποιοι τις παρέχουν ε, θελοντικά και ε, το πρόβλημα είναι ότι οι καταναλωτέ νιώθουν ότι του παραπλανούν αν δεν είναι διαθέσιμες αμέσω. Πολλοί λένε ότι τα προϊόντα είναι πολύ ακριβά, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πάντα χρησιμοποιεί αυτό το επιχείρημα, ενώ η έκθεση τη ίδια τη επιτροπή λέει ότι ίσω ο κλάδο μπορεί να υπερέβαλε όσον αφορά το κόστο τη ε, αναγραφή. Μπορεί να γίνει για διάφορους λόγους. Ε, μπορεί να είναι για θέματα ευημερία των ζώων, για περιβαλλοντικούς λόγους ή γιατί προτιμούν ε, ντόπια εγχώρια προϊόντα. Ε, δεν φαίνεται να είναι λογικό για μένα να υπάρχει αναγραφή για τα περισσότερα νοπάκρο κρέατα του τόπου προέλευσης και όχι για όλα. Όσον αφορά το κρέας αλόγου, ήδη υπάρχει ε, σύστημα εχνηλασιμότητας και δεν καταλαβαίνω πού βρίσκεται το πρόβλημα. Τελικά θέλουμε απλώς να διασφαλίσουμε ότι οι καταναλωτές γνωρίζουν από πού προέρχεται το κρέας που καταναλώνουν, ε, μπορούν να έχουν εμπιστοσύνη στην αλυσίδα διαμονή, διανομής και μπορούν να δώσουν στους καταναλωτές αυτό που ζητούν. μπορουν να εχουν εμπιστοσυνη στην αλυσιδα διανομη διανομης τέτοιο, έχουν δικαίωμα να τους δίνονται αυτές οι πληροφορίες και εμείς πρέπει να διασφαλίσουμε ότι θα τις λάβουν. Ευχαριστώ πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Η κυρία Γιατανμάκη. Ευχαριστώ πολύ. Θα είμαι πολύ σύντομη. Θα ήθελα να τονίσω τη διαφάνεια και το δικαίωμα των καταναλωτών να είναι σωστά ενημερωμένοι σχετικά με την ε, χώρα καταγωγής ή τον τόπο προέλευσης ε, για κάποια τρόφιμα. Ταυτόχρονα πρέπει να γνωρίζουμε ότι οι απαιτήσει αυτές ε, μπορεί να είναι δαπανηρές ε, για τον σχετικό τομέα. Θα πρέπει λοιπόν το διοικητικό άχθος ε, να κατανεμηθεί ίσα χωρίς να στρεβλώνεται ο ανταγωνισμός. Ε, αλλά τα νούμερα που έχω δει μέχρι τώρα είναι πολύ ψηλά όσον αφορά τις δαπάνες δεν θα πρέπει να είναι εύκολο ε, για τον ε, τομέα να κρύβεται πίσω από ε, κακές διατάξεις και να αναλαμβάνεται δράση μόνο αναδρομικά σε περίπτωση που κάτι πάει στραβά. Θα πρέπει δηλαδή, αν συμβεί οτιδήποτε, να μπορούν να μας ενημερώσουν ήδη την επόμενη μέρα από πού προέρχεται η συγκεκριμένη τροφή. είμαι δηλαδή υπέρ της υποχρεωτικής επισήμανσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Μπόιλαν δεν είναι παρούσα. Η κυρία Ριβάζη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Εγώ από την άλλη έχω κάποιες απο... Ε, κάποια ερωτήματα που θέλω να θέσω στην Κομισιόν γιατί δεν καταλαβαίνω την αλλη εχω καποιες καποια ερωτηματα που θελω να θεσω στην κομισιον γιατι δεν καταλαβαινω την συμπεριφορα τους. Έχουμε μια έκθεση ε, το Δεκέμβριο του 2013 που μας λέει ότι είναι απαραίτητο να αναγράφεται ε, η προέλευση στα κτηνοτροφικά πρόγραμμα. Στι 25 του 2015 έχουμε μια νέα έκθεση στην οποία μας λέει ότι πρέπει να υπογράφεται υποχρεωτικά η προέλευση για τα γαλοκτοκομικά. Έχουμε τους καταναλωτές οι οποίοι επιθυμούν να γνωρίζουν την προέλευση, την καταγωγή των τροφίμων τους. Και τι κάνει η Κομισιόν, τίποτα. Δεν έχει έρθει η στιγμή να κινητοποιηθείτε. Μέχρι στιγμής η προτεραιότητα ήταν στα ε, καλακτοκομικά, στο τύρι, ε, αργότερα στο κρέας και μας λέτε ότι θα κοστίσει ακριβά. Μα όχι, στην Γαλλία το εφαρμόζουμε. Ήδη ε, όλοι επωφελούνται. Επωφελούνται οι καταναλωτέ που γνωρίζουν τι είναι αυτό που τρώνε. Επωφελούνται οι παραγωγοί γιατί μπορεί ο καταναλωτή να επιλέγει το προϊόν του. Επομένω έχει έρθει και έχει περάσει ο καιρό που θα έπρεπε η Κομισιόν να έχει κινητοποιηθεί. Υπάρχει επίσης το ζήτημα της, του δικαιώματος που έχει ο καταναλωτής να γνωρίζει όχι μόνο από που προέρχεται, αλλά επίσης, από ποια χώρα, αλλά επίσης να γνωρίζει για παράδειγμα εάν τα ζώα από τα οποία προέρχεται το τρόφιμο του, το, τα κρέατα ή τα γαλακτοκομικά, έχει τραφεί έχει ε, ε, με χρήση ζωοτροφών που προέρχονται από ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Υπάρχει επίσης και ένα ζήτημα του περιβάλλοντος. Αυτή τη στιγμή στην, το, γάλα που έρχεται από τη Δανία στη Γαλλία είναι πιο φτηνό από το γαλλικό γάλα. Γιατί, Γιατί δεν αξιοποιούμε τα συστήματα μεταφορέ που θα έπρεπε. Είναι, υπάρχει και μια περιβαλλοντική διάσταση λοιπόν σε αυτό, στι εκπομπέ του διοξιδίου του άνθρακα για τη μεταφορά αυτών των ε, ε τροφίμων. Θα έπρεπε λοιπόν να δώσουμε τον, στον καταναλωτή το δικαίωμα, τη δυνατότητα να κάνει τις επιλογές του με βάση τις αρχές του και με αυτόν τον τρόπο να καταπολεμήσουμε ε, και τη, ε, να βοηθήσουμε και τη βιοποικιλότητα για να καταπολεμήσουμε και πρακτικές κτηνοτροφικές που δεν θέλουμε. Και διαπιστώνουμε ότι είναι η Κομισιόν η οποία την μπλοκάρει αυτές τις πρωτοβουλίες. Ευχαριστώ πολύ, ο κύριος Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η θέση της ομάδας μας είναι οι σχέσεις ε, που έχουν να κάνουν με την αναγραφή για όλα τα προϊόντα τα οποία δεν περιλαμβάνονται στην υποχρεωτική αναγραφή του τόπου προέλευσης. Εμείς θέλουμε να είναι υποχρεωτική και για όλα τα προϊόντα της Ένωσης. Βέβαια η υποχρεωτική αναγραφή δεν διασφαλίζει την ποιότητα ε, του προϊόντος, ε, αλλά επιτρέπει τουλάχιστον στους καταναλωτές να επιλέγουν συνειδητά το κρέα τους, ε, τα μακαρόνια τους, τη ζάχαρή τους, όλα τα προϊόντα τα οποία παράγονται στις περιοχές μας. Είναι αλήθεια βέβαια ότι δεν μπορούμε να έχουμε την απέτηση να φτάσουμε σε αυτό το προϊόν από τη μια στιγμή στην άλλη. Πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα σε επιχειρήσεις και στου παραγωγού να προσαρμοστούν στην νομοθεσία και να φροντίσουν η παραγωγή τους να είναι αντίστοιχη. Είμαστε λοιπόν σε ένα μεταβατικό στάδιο, διότι αφενό ε, οι παραγωγοί θα επιλέξουν ε, να υπάρχει αναγραφή του τόπου προέλευση, ενώ κάποιοι θα επιλέξουν να μην το κάνουν. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει την υποχρέωση να φροντίσει όσοι επιλέξουν να υπάρχει αναγραφή της, ε, του τόπου προέλευσης θα έχει και μια προστιθέμενη αξία λόγω της αναγραφής αυτής. Ενώ όσοι επιλέξουν να μην το κάνουν δεν θα πρέπει με κανένα τρόπο να αναφέρονται στην προέλευση των προϊόντων ε, και να οδηγήσουν έτσι σε αθέμητο ανταγωνισμό. Και αναρωτιέμαι γιατί επιλέξατε να μην ε, ρυθμίσετε αυτά τα εθελοντικά προγράμματα όπως έγινε στο παρελθόν με τις ε, ε γεωγραφικές ενδείξεις και με τα προϊόντα. Αυτή τη στιγμή η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λέει ότι όταν ε, αναγράφεται, δεν θα πρέπει να ε, υπάρχει παραπλανητικό στοιχείο για τον τόπο προέλευσης ή τη χώρα καταγωγής, αλλά οι αρμόδιες αρχές είναι αυτές οι οποίες θα εφαρμόσουν τη συγκεκριμένη αρχή και οι αρμόδιες αρχές δεν είναι ε, άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν συμφέρον γιατί περασπίζονται τα εθνικά συμφέροντα. Ποιο είναι λοιπόν αυτός ο οποίος προασπίζεται τα συμφέροντα της εσωτερικής μας αγοράς και ποιο προστατεύει τα προϊόντα μας όταν πολλούνται εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ η κυρία Σαλβίνη δεν είναι εδώ. Επομένως θα ξεκινήσουμε με τους υπόλοιπους ομιλητές, ε, η κυρία Σόμερ. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Το θέμα της αναγραφής της χώρας καταγωγής είναι ένα θέμα που μας απασχολεί εδώ και πολλά χρόνια. Σχετίζεται με τον κανονισμό για την ε, ενημέρωση σχετικά με τα τρόφιμα και Είμαστε αρκετοί αυτοί που συμμετείχαν στις διαπραγματεύσεις κατά την προηγούμενη θητεία. Το Συμβούλιο, το αίτημα του Κοινοβουλίου, το ενέκρινε μόνο υπό την προϋπόθεση να πραγματοποιούνται μελέτες αντικτύπου. Αυτό έγινε από την Κομισιόν. Αλλά και πρόσφατα ακόμα είδαμε ότι η Κομισιόν απορρίπτει το σχέδιο ψηφίσματος. Είναι διαφορετική η πολιτική βούληση. Στην περίπτωση αυτή δεν χρειάζεται να ε, αναθέτει μελέτες αντικτύπου η Κομισιόν. Διαπίστωσε ότι το κόστος είναι υπερβολικό ιδιαίτερα όσον αφορά το κρέας ε, στα μεταποιημένα τρόφιμα. Εδώ απέριψε υποχρεωτική αναγραφή, ενώ για το ε, γάλα, γαλακτοκομικά και άλλα είδη κρέατος ε, η Κομισιόν κατέληξε στο συμπέρασμα ότι το κόστος δεν ανταποκρίνεται στο όφελος ο καταναλωτής δεν είναι διατεθειμένος να πληρώσει περισσότερα για την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής. Γι' αυτό η Κομισιόν δεν έχει προγραμματίσει νομοθετική πράξη και αυτό το γνωρίζουμε αρκετό καιρό. Στο νέο σχέδιο ψηφίσματος που έχουμε, στη νέα αυτή προσπάθεια, γίνεται προσπάθεια να πείσουμε την Κομισιόν να υπάρχει υποχρεωτική αναγραφή για τα ελαφρώς μεταποιημένα τρόφιμα, ε, για το κρέας και για τα γαλακτοκομικά. Και η Κομισιόν διαπιστώνει ότι όντως αυξάνεται το κόστος ανάλογα με τον βαθμό μεταποίησης των τροφίμων Όσο περισσότερο μεταποιημένο είναι ένα προϊόν, ε, τόσο αυξάνεται το κόστος αναγραφής ε, της προέλευσης των τροφίμων, των συστατικών του. Το πρόβλημα όμως εδώ είναι ακριβώς αυτός ο όρος, ε, τα ελαφρώς μεταποιημένα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένος ορισμός. την συζήτηση αυτή σχετικά με το τι είναι ελαφρώς μεταποιημένο, τι είναι πιο μεταποιημένο κλπ. Είναι μια συζήτηση την οποία είχαμε κατά τις διαπραγματεύσεις ε, για τον ε, κανονισμό ε, για την ενημέρωση σχετικά με τα τρόφιμα και διαπιστώσαμε ότι δεν είναι δυνατόν να γίνεται έτσι η αναγραφή. Γι' αυτό Βρίσκω και λάθος την πρόταση. Ε, τα αλλαντικά, ένα λουκάνικο δεν είναι ελαφρώς μεταποιημένο, δεν θα πιστέψετε τι περιέχει. Υπάρχουν πολλά βήματα μεταποίησης μέχρι να γίνει λουκάνικο. Και δεν είναι και όλα τα λουκάνικα ίδια που θα βάλουμε τα όρια λοιπόν. Θα ήθελα να προτείνω να ζητάμε τουλάχιστον έναν ορισμό. και υπάρχει το όνομά μου εδώ πέρα ως ε, συνεισηγήτρια. Ε, χαίρομαι λοιπόν που ε, έχετε αφήσει στο σχέδιο ψηφίσματος το αίτημα για ορισμό. Το θέμα αυτό σχετίζεται και με την προφορική ερώτηση. Είναι βασική αρχή του δικαίου ότι όλα θα πρέπει να έχουν κάποιον ορισμό. Όταν διαπιστώσουμε αν μπορούμε να έχουμε ορισμό, θα ε, διαπιστώσουμε αν μπορούμε να έχουμε υποχρεωτική αναγραφή, διότι αν δεν μπορούμε να έχουμε ορισμό για, τα, για την κατηγορία αυτή των προϊόντων, τότε δεν θα μπορούμε να έχουμε και σχετικό κανόνα. Ε, άλλο πρόβλημα είναι ότι δεν περιμένουμε την απάντηση στην προφορική ερώτηση. προς την Κομισιόν. Λέμε, σας παρακαλώ εξετάστε το θέμα αυτό, αλλά θέλουμε ε, την υποχρεωτική αναγραφή για τα ε, ελαφρώς μεταποιημένα προϊόντα με κρέας και γαλακτοκομικά γι' αυτό. Βρίσκω λάθος το να υποβάλουμε το κείμενο του ψηφίσματος ως έχει και γι' αυτό. Έχω αφαιρέσει και την υπογραφή μου από το κείμενο του ψηφίσματος, ενώ παραμένει στην προφορική ερώτηση. Επίσης, αν τα αποτελέσματα της μελέτης αντικτύπου της ε, Κομισιόν ε, δεν βολεύουν τους συναδέρφους, ε, τότε την κατηγορούμε ότι ότι προδικάζει τα αποτελέσματα. Αλλά εγώ έχω απόλυτη εμπιστοσύνη στην Κομισιόν. Υπάρχουν και διάφορες γενικές διευθύνσεις που ασχολούνται με το θέμα αυτό. Εάν λέμε ότι δεν ισχύουν αυτά που γράφει η Κομισιόν, τότε ας μην κάνει και τη δουλειά όλοι. Δεν μπορούμε να δίνουμε τέτοια απάντηση ανάλογα με την ατζέντα του κάθε κόμματο. Επίσης, βρίσκω λάθος να ε, γίνουν πιο ακριβά κάποια βασικά τρόφιμα ε, για ανθρώπους που πιθανότατα δεν θα ενδιαφέρονται καν για την χώρα καταγωγής. Και ένα τελευταίο σημείο που επίσης ε, πάντα ε, μου προκαλεί κάποια δυσαρέσκεια είναι η συσχέτιση του θέματος αυτού με τα σκάνδαλα στον τομέα των τροφίμων. Άλλωστε το σκάνδαλο με το αλογίσιο κρέας δεν θα το είχαμε αποτρέψει με την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής. και το θέμα τη επισήμανση των τροφίμων ε, δεν μπορούμε πάντα να το συσχετίζουμε με την ασφάλεια των τροφίμων. Συχνά υπάρχουν πολύ σημαντικοί εθνικοί λόγοι για κάποιες ε, διατάξεις. Είμαι απολύτως πεπισμένη ότι ε, κρύβεται πολύ προτεξιονισμός πίσω από όλα ε, αυτά τα αιτήματα. Δεν θα ήθελα να τα στηρίξω λοιπόν. Σας ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Ο κύριος Παχνιό. Και εγώ, όπως η συναδελφός μου, θέλω να απευθυνθώ στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Γιατί. Πρώτον, Νομίζω ότι όλοι το έχουμε αντιληφθεί και είναι και ο λόγος που θέλουμε να υποστηρίξουμε αυτό το ψήφισμα είναι ότι τρία χρόνια μετά από το σκάνδαλο, το διατροφικό σκάνδαλο του κρέατος αλόγου συνεχίζουμε να μην μπορούμε να ικανοποιήσουμε το 70% των τονίζων των Ευρωπαίων καταναλωτών οι οποίοι απαιτούν να αναγράφεται η προέλευση της ε, του κρέατος που χρησιμοποιείται σε ε, ε, έτοιμα ε, προμαγειρεμένα ε, τρόφιμα. Γι' αυτό είχαμε ζητήσει από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να επιταχύνει την αναθεώρηση του κανονισμού ε, που αφορά τα δικαιώματα του καταναλωτή στην ενημέρωσή του, έτσι ώστε να μπορεί να γνωρίζει ο καταναλωτή από πού έχουν προέλθει τα συστατικά αυτών των μεταπημένων τροφίμων. Και η απάντηση της Κομισιόν ήταν ουσιαστικά μία έκθεση, η έκθεση του 2013 που αναφέρθηκε, ε, που αξιολογεί το κόστος που θα είχε η υποχρεωτική αναγραφή. Και λέει ότι το κόστος θα ήταν υπερβολικό για την βιομηχανία τροφίμων και για τους καταναλωτές. Η εκτιμά μια αύξηση της τάξης του 20% στις τιμές αυτών των τροφίμων. Πιστεύω ότι το πρόβλημα είναι εδώ, στην πραγματικότητα. Ότι ασκείται ισχυρή πίεση. Ότι αυτό που απασχολεί ορισμένους που ασκούν αυτήν την πίεση δεν είναι τα, ο αντίκτυπος στους καταναλωτές και στο γεγονό ότι οι καταναλωτές δεν γνωρίζουν τι τρώνε, αλλά το κόστος που θα είχε για τη βιομηχανία τροφίμων. Εγώ όμως κρίνω ότι στην πραγματικότητα ε, αυτό το, το κόστος το έχουμε υπερεκτιμήσει. Άλλες μελέτες έχουν ε, αποδείξει ότι η αύξηση στην κατανάλωση των μεταπημένων τροφίμων με βάση το κρέας ήταν πολύ μικρή, ανεξαρτήτως. Ε, της υποχρέωσης αναγραφής της ε, της προέλευσης. Και αυτό το έκαναν συγκρίνοντας ε, την περίπτωση ε, τροφίμων τα οποία είχαν βάσει το κρέας και άρα ήταν υποχρεωτική ανατροφή, ε, αναγραφή με βάση άλλα τρόφιμα που δεν, τα οποία δεν ήταν. Άρα δεν είναι σωστά τα στοιχεία της Κομισιόν. Μέχρι και σήμερα το 50% των ε, τροφίμων που περιέχουν ε, ε, προϊόντα κρέατος δεν το αναφέρουν. 65% των μεταποιημένων τροφίμων με κατόπουλο δεν αναφέρουν την προέλευση Και τα λοιπά. Επομένως χρειάζεται να συνεχίσουμε την πολιτική πίεση προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το ψήφισμα είναι μία μέθοδος πολιτικής πίεσης έτσι ώστε η αναγραφή της προέλευσης να γίνει υποχρεωτική. Όπως το αναφέρει και ο εισηγητής της, η διαφάνεια ε, θα πρέπει να εφαρμόζεται και στο, στα γαλακτοκομικά και στο κρέας και στο κοτόπουλο κτλ. Η, στη, στη, στη, στη, η Γαλλία είναι ένα από τα κράτη-μέλη που ζητούν να γίνει κάτι τέτοιο για τα γαλακτοκομικά και πολλά άλλα κράτη-μέλη και πολλοί Ευρωπαίοι πολίτες ζητούν την υποχρεωτική αναγραφή. Ο Πρόεδρος. Κύριοι συνάδελφοι, δέκα ευρωβουλευτές έχουν ζητήσει το λόγο, γι' αυτό θα σας ζητήσω όσο μπορείτε να είστε στο δυνατόν πιο σύντομοι στις παρεμβάσεις σας. Κύριε Γκροστέτ, ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Υπάρχουν οι έρευνε του Ευρωβαρομέτρου που παρεπιπτόντω αναφέρονται και στο κείμενο και αποδεικνύουν ότι από πλευρά καταναλωτών υπάρχει πραγματικά αίτημα να γνωρίζουν από πού προέρχονται και ποια είναι η προέλευση αυτών των προϊόντων που ε, φτάνουν στο πιάτο τους. Ε, αυτή η αναγραφή λοιπόν του τόπου προέλευσης μου φαίνεται σημαντική γιατί μπορούμε να διαφοροποιήσουμε τα προϊόντα και να ε, προσδώσουμε αξία, σαν διαφήμιση ας πούμε, την προέλευση ενός προϊόντων. Το πρόβλημα του κόστους είναι ένα πρόβλημα το οποίο αναφέρουν όλοι. Νομίζω ότι εάν είναι ε, προαιρετική η αναγραφή του τόπου προέλευσης, τότε εκεί θα υπάρχει θέμα κόστος, γιατί κάποια προϊόντα θα είναι πιο ακριβά από κάποια άλλα και αυτό θα δημιουργήσει πραγματική διαφορά. Εάν ε, η αναγραφή του τόπου προέλευσης είναι υποχρεωτική, ε, τους αφορά όλους, οπότε όλοι αναλαμβάνουν το κόστος με, με τον ίδιο τρόπο και δεν υπάρχει πλέον καμία διαφοροποίηση. Στην πραγματικότητα, για αυτό το θέμα του κόστους υπάρχουν κάποιες μελέτες οι οποίες ε, είναι εκ διαμέτρου αντίθετες. Κάποιες λένε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπερέβαλε ως προς το κόστος. Εγώ πραγματικά θα ήθελα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τα επανεξετάσει όλα αυτά σοβαρά ε, με ακρίβεια και να μας πει τι ακριβώς συμβαίνει. Διότι είναι πολύ μεγάλες οι αποκλήσεις μεταξύ των διαφόρων μελετών ε, και τα στοιχεία είναι τελείως ε, διαφορετικά. Πώς μπορούμε λοιπόν να βασιστούμε στα συμπεράσματα αυτής της της κάθε μελέτης. Ε, θα καταθέσω και τροπολογίες με την κυρία Ντελαέ προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριο Σουητέμα. Ναι, ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε έχω και εγώ κάποιες ερωτήσεις ε, για το ψήφισμα αυτό. Πρώτον, το ανέφερε και η κυρία Σόμερ, πώς μπορούμε να έχουμε ένα σαφή ορισμό. Ποια είναι η διαφορά μεταξύ ελαφρής μεταποίησης και ε, υψηλής μεταποίησης. Ε, πρέπει να υπάρξει ένας ορισμός να το διευκρινίσουμε αυτό και μετά να μιλήσουμε για την ε, αναγραφή. Και πρέπει να σκεφτούμε τι θέλουν οι καταναλωτές. Το πρώτο πράγμα που αφορά τους καταναλωτές κατά την άποψή μου είναι η τιμή, η γεύση, μετά η ημερομηνία λήξεως και στο τέλος ίσως ο τόπος προέλευσης ή η χώρα καταγωγής εύκολα μπορούμε να κάνουμε νέα νομοθεσία, αλλά συχνά δεν σκεφτόμαστε πώς μπορούν οι παραγωγοί να ε, κερδίσουν όσα ε, δαπανούν ε, λόγω της υψηλής γραφειοκρατίας. Θα πρέπει να στραθούμε και σε αυτό. Και επίση, γιατί θέλουμε να έχουμε υποχρεωτική αναγραφή σε επίπεδο κράτου μέλου. Το Κοινοβούλιο, ω νομοθέτης ε, ε, καταρτίζει ευρωπαϊκή νομοθεσία που θα έπρεπε να ισχύει για όλα τα κράτη-μέλη. Γιατί να υπάρχει λοιπόν διαφοροποίηση στην υποχρεωτική αναγραφή σε επίπεδο κράτου μέλου και να μην υπάρχει ένα πρώτο βήμα. Να υπάρχει μια ευρωπαϊκή ε, ετικέτα ή μια μη ευρωπαϊκή ετικέτα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ολοκληρώνει το κατάλογο των ομιλητών, γιατί αλλιώς ε, όλο θα προσθέτουμε ονόματα. Ο κύριος Χέλνερ. Ευχαριστώ πολύ. Συμφωνώ με τους προλαλήσαντες σε ένα σημείο. Δεν καταλαβαίνω ποιο είναι το πρόβλημα. Εγώ θα το έλεγα αντίστροφα. Άκουσα ότι οι καταναλωτές το θέλουν. Ε, πολλοί παραγωγοί ήδη ε, παρέχουν τη δυνατότητα αυτή. Δηλαδή αυτοί που θέλουν μπορούν να το έχουν, αυτοί που δεν θέλουν να πληρώσουν για κάτι τέτοιο δεν χρειάζεται να πληρώσουν για κάτι τέτοιο. Εάν όλοι οι καταναλωτές το θέλανε τόσο πολύ, θέλανε τόσο πολύ την υποχρεωτική αναγραφή, τότε και όλη η παραγωγή ε, θα ανέγραφαν ε, την χώρα καταγωγής. Γιατί να θέλει κανείς υποχρεωτική αναγραφή για λόγους ε, καλής μεταχείρισης των ζώων, προστασία του περιβάλλοντος κλπ. Δεν ξέρω, αλλά τελευταία φορά που θυμάμαι εγώ, στην Επιτροπή μας θέλαμε κοινού κανόνες για να έχουμε κοινή αγορά με κοινά πρότυπα. Εκαταλείψατε την ιδέα, εγώ όχι. Και η τελευταία μου παρατήρηση. Θέλουμε υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής. Έτσι μήπως κάνουμε πιο σημαντικά τα σύνορα στην ε, Ευρώπη. Ίσως να μην είναι οι ευρωσκεπτικιστές ε, η απειλή στην Ευρώπη, ίσως να είναι η νέα νομοθεσία η απειλή. Αλλά σε μια Ευρώπη των περιφερειών, γιατί να αναφέρουμε την χώρα καταγωγής ε, και να μην λέμε ότι κάτι προέρχεται από τη Φλάνδρα, την Βαβαρία, το Σκόνε στη Σουηδία. Θα λέγατε ότι δεν είναι πρακτικό. Μπορεί να πείτε ότι δεν μας ενδιαφέρει κιόλας. Θα σας πω όμως κάτι και η πρότασή σας ε, δεν ε, έχει πολύ πρακτική βάση. Πιθανότατα να είναι και αδύνατο να πραγματοποιηθεί. Thank you very much. Ευχαριστώ κύριο Σορνάνο. Ε, Ευχαριστώ. Ένα χρόνο πριν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όταν συζητούσαμε το ζήτημα των ετικετών της ετικετοθεσίας η οποία εξαπατούσε τον καταναλωτή μας έλεγε ότι δεν θα έπρεπε, δεν επιτρέπεται η εξαπάτηση του καταναλωτή αναγράφοντας ψευδή προέλευση του τροφίμου. Επίσης, για τα προϊόντα κρέατος υπάρχει μεγάλη, είναι πολύ σημαντικό για τον καταναλωτή να γνωρίζει από πού προέρχονται. Αυτή η πρόταση λοιπόν που θα ε, κάνει υποχρεωτική την αναγραφή και για τα μεταποιημένα τρόφιμα προστίθεται σε μια συζήτηση που κάνουμε εδώ και τρία χρόνια η οποία ξεκίνησε με το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου στα λαζάνια. Τα επιχειρήματα είναι ξεκάθαρα. Είναι γνωστό ότι ορισμένες ε, επιχειρήσεις έχουν επιδιώξει να μας πείσουν ότι το κόστος της υποχρεωτικής αναγραφής θα είναι πολύ υψηλό. Ωστόσο οι καταναλωτές το επιθυμούν για λόγους διαφάνειας. Το γεγονό ότι δεν υπάρχει αυτή η ε, προσέγγιση στην πραγματικότητα δημιουργεί ε, άνισο ανταγωνισμό με, αναμεταξύ των επιχειρήσεων που δραστηριοποιούνται στην ευρωπαϊκή αγορά. Πιστεύω λοιπόν ότι το ζήτημα αυτό οφείλει να μα απασχολήσει μέσω του, του, και μέσω της που θα ακολουθήσει. Ευχαριστούμε κύριε Ντόρφμαν. Ευχαριστώ. Ναι, στην Ευρώπη έχουμε προϊόντα με αναγραφή της χώρας καταγωγής, η οποία ελέγχεται κιόλας. Κατόπιν έχει κανείς την δυνατότητα από μόνος του κάποιος να αναγράφει την χώρα καταγωγής και θα μπορούσαμε να έχουμε εδώ βελτιώσεις. Πιστεύουμε ότι θα ήταν λογικό να έχουμε πιο ακριβείς κανόνες σχετικά με αυτήν την προαιρετική ανάγραφη, ώστε να ελέγχεται ε, η ακρίβεια των ε, στοιχείων αυτών. Και κατόπιν έχουμε τα προϊόντα όπου δεν υπάρχει αναγραφή της χώρας καταγωγής. Γιατί πρέπει εμείς πάντα να λέμε στον καταναλωτή τι πρέπει να κάνει. Το ερώτημα αυτό δεν συνδέεται καθόλου με την ασφάλεια των τροφίμων. Είτε ένα προϊόν προέρχεται από την Ιταλία, την Αυστρία ή τη Γαλλία ή τη Σουηδία. Δεν έχει να κάνει με το αν είναι ασφαλέ. Πρέπει όλα να είναι ασφαλή. Και αν δεν είναι ασφαλή τα τρόφιμα, τότε έχουμε ένα πολύ πιο βασικό πρόβλημα στην Ευρώπη. Και βέβαια μπορεί κανείς να μιλήσει για τα προϊόντα όπου είναι προαιρετική αναγραφή, είναι πιο ακριβά και γι' αυτό θα πρέπει να προωθήσουμε τα τρόφιμα αυτά αυξάνοντας τη τιμή και σε όλα τα υπόλοιπα τρόφιμα. Αγαπητοί συνάδελφοι, όμως ε, δεν, δεν παίρνουν ε, όλοι οι πολίτες ε, της Ευρώπης τον ίδιο μισθό με εμάς. Υπάρχουν καταναλωτές στην Ευρώπη που εξετάζουν πολύ προσεκτικά τι θα αγοράσουν όταν πηγαίνουν για ε, ψώνια στο σούπερ μάρκετ. Θα πρέπει λοιπόν ε, να σκεφτούμε πράγματι αυτό. Θέλουμε να πούμε ότι θα ε, ενισχύσουμε την προαιρετική αναγραφή στα τρόφιμα και ότι οι παραγωγοί θα θέλουν κατόπιν να, κάνουν να έχουν αναγραφή της χώρας καταγωγής. Τώρα, το εάν σε όλα τα γιαούρθια και τυριά της Ευρώπης και τα λουκάνικα, ε, εάν ε, σε όλα αυτά αναγράφεται ε, από πού προέρχονται δεν νομίζω ότι θα αλλάξει τίποτα στην αγορά. Οι πωλήσει δεν θα αυξηθούν ή θα μειωθούν αν ξέρουμε ότι το λουκάνικο αυτό προέρχεται από την Ουγγαρία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ήθελα και εγώ να πω την άποψή μου για το θέμα αυτό και να σας πω ότι τουλάχιστον τα στοιχεία που γνωρίζω εγώ και τα στατιστικά στοιχεία ε, που έχω στη διάθεσή μου λένε ότι ο καταναλωτής ε, προσέχει την ε, προέλευση όταν πρόκειται για νοπά κρέατα, όχι τόσο για τα μεταποιημένα κρέατα. Ε, τους ενδιαφέρει περισσότερο η συνταγή, η παράδοση, η καινοτομία και η δημιουργικότητα πράγματι βλέπει με θετικό μάτι την αναγραφή του τόπου προέλευσης, αλλά όχι τόσο ουσιαστικά όπως ε, στην περίπτωση της προέλευσης του νοπού κρέατος. Κυρίως ε, ε, επαναλαμβάνω με βάση τα στοιχεία που έχω εγώ στη διάθεσή μου. Δεν μπορούμε να χρησιμοποιούμε το επιχείρημα της ποιότητας και της ασφάλειας των τροφίμων για να Υπεραμεινθούμε τις θέσεις ότι είναι υποχρεωτική η αναγραφή του τόπου προέλευσης του κρέατος στο μεταποιημένο προϊόν, διότι είναι σαν να ε, ε, αμφισβητούμε αυτή τη στιγμή το σύστημα εγγυήσεων της διατροφικής αλυσίδας που έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση και εγώ το εμπιστεύομαι το σύστημα. Επομένως, δεν θεωρώ ότι ε, αποτελεί λογικό επιχείρημα το, ο ισχυρισμός ότι προσθέτει ασφάλεια και ποιότητα. Ε, διότι αλλιώς αμφισβητούμε αυτή τη στιγμή αυτά τα οποία συμβαίνουν. Ε, πράγματι είναι σημαντικό το κόστος και το είπανε κάποιες συνάδελφοι, το κόστος είναι πάρα πολύ σημαντικό για τον κλάδο αλλά και για τους καταναλωτές και είναι κάτι το οποίο πρέπει να προσέξουμε. Ε, σαφώς και μας ενδιαφέρει η υγεία, το περιβάλλον και σίγουρα η οικονομική κατάσταση των καταναλωτών. Εμείς ε, δεν θεωρούμε ότι, είναι, ε, θεωρούμε ότι είναι ένα προστατευτικό μέτρο και μέτρο επανεθνικοποίησης, διότι οι καταναλωτές ε, το βλέπουν με θετικό μάτι και είναι προαιρετικό, επομένως τι πρόβλημα υπάρχει θα μπορούσαμε να το δεχτούμε. Εγώ θεωρώ ότι είναι σαφέστατα μέτρο προστατευτισμού και εθνικοποίησης και θα ήθελα να επενθυμίσω το εξή. και το λέω και στα μέλη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. ο ΠΟΕ ήδη έχει γνωμοδοτήσει κατά της ε, παρανομίας ε, της υποχρεωτικής αναγραφής ε, του τόπου προέλευσης στις Ηνωμένε Πολιτείες και χρειάστηκε να το καταργήσουν. Αυτή είναι λοιπόν γνωμοδότηση του ΠΟΕ, ο οποίος γνωμοδότησε για την νομιμότητα ενός αντίστοιχου συστήματος με αυτό το οποίο προσπαθούμε να εφαρμόσουμε στην Ευρώπη. Οι Ηνωμένε Πολιτείε λοιπόν ε, κατήργησαν το σύστημα και σας το λέω αυτό προκειμένου να λάβουμε υπόψη μας όλες τις παραμέτρους. Ε, δεν ξέρω ε, και ο ΠΟΕ μπορεί να έχει άποψη. Πολλά πράγματα λοιπόν είναι αποφάσεις που ίσως δεν μου αρέσουν, αλλά αυτές είναι αποφάσεις που πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. Εάν λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι προαιρετικό, ε, ποιος λόγος υπάρχει να προσθέσουμε κάτι παραπάνω. Δεν καταλαβαίνω την πρωτοβουλία για ποιο λόγο γίνεται και γι' αυτό και είμαι κατά. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κέστιγκερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Η κυρία Σόμερ μάλλον γνωρίζει γιατί δεν λειτουργεί το μικρόφωνο μου. Μετά τις διαφορετικές παρεμβάσεις που ακούσαμε, ε, θα ήθελα εγώ να υποστηρίξω την υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής. Θέλουμε διαφάνεια. Πολλοί καταναλωτές προτιμούν τρόφιμα, ιδιαίτερα προϊόντα κρέατος, ε, με αναγραφή του τόπου προέλευσης και γενικά οι επιχειρήσεις ε, στην Ευρώπη πρέπει να πληρούν πολλές προϋποθέσεις κατά την παραγωγή. Ε, <clears throat> αναφέρομαι ιδιαίτερα στα μεταποιημένα προϊόντα κρέατος, όπου συχνά βλέπουμε πολλές καταχρήσεις και νομίζω ότι θα ήταν πολύ χρήσιμο να σκεφτούμε περαιτέρω την υποχρεωτική αναγραφή και θα ήταν ενδιαφέρον νομίζω και για την Κομισιόν να εξετάσει την, ε, ε, την εφαρμογή της νομοθεσίας αυτής και στα αυγά και τα προϊόντα αυγών. Έχουμε πολλά εισαγόμενα αυγά από τρίτες χώρες, από την Ουκρανία για παράδειγμα, και σε πολλά προϊόντα μέσα, σε ζυμαρικά κλπ. Και θα ήθελα να αναφέρω άλλη μία πτυχή. Αυτή τη στιγμή συζητάμε σε υψηλού τόνου στην Ευρώπη την ε, εμπορική συμφωνία με τις Ηνωμένε Πολιτείε. Αλλά όσον αφορά τις τρίτες χώρες ε, δεν υπάρχει καθόλου ηχνηλασιμότητα. Πιστεύω λοιπόν ότι θα ήταν προ συμφέρον του Ευρωπαίου παραγωγού και θα ήταν υπέρ της διαφάνειας να έχουμε η υποχρεωτική αναγραφή της χώρας καταγωγής. Ευχαριστώ. κυρία Καμπεθόνου Ρουίς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Λοιπόν, εγώ καταρχάς ε, θα ήθελα να πω ότι εγώ δεν έχω καμία αμφιβολία ότι το πρόβλημα ε, μπορεί να λυθεί, ότι η ετικέτα μπορεί να αυξήσει τόσο πολύ το κόστος ενός προϊόντων και το να προσθέσουμε ένα στοιχείο θα αυξήσει τόσο πολύ το κόστος. Ε, αυτός ο οποίος παράγει και πουλά πραγματικά ε, καθορίζει μια τιμή με βάση το προϊόν το οποίο σκοπεύει να πουλήσει και σε ποιον απευθύνεται. Εγώ νομίζω ότι τα πράγματα είναι αντίθετα και τη γνωρίζουμε όλη αυτή την αρχή της κοστολόγησης και της τιμολόγησης ενός προϊόντων. Λοιπόν, δεν θεωρώ ότι αυξάνεται τόσο πολύ η τιμή ενός προϊόντων και μάλιστα ε, τόσο μεγάλη αύξηση. Αμφισβητώ λοιπόν το κατά πόσον είναι θέμα τιμή μόνο και αφού είναι προαιρετικό γιατί υπάρχει τόσο πρόβλημα. Θεωρώ ότι φέρπουν και άλλοι λόγοι και θα ήθελα να μου πείτε ποιοι είναι αυτοί. Έχουν γίνει μελέτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για την τιμή και πραγματικά θα ήθελα να ξέρω αν υπάρχουν άλλοι λόγοι που θα μπορούσαν να ε, δημιουργήσει πρόβλημα. Μπορεί οι παραγωγοί ε, να έχουν πρόβλημα για άλλο λόγο για να μας πούν από πού προέρχονται τα προϊόντα. Νομίζω ότι έχει σαφή σχέση με την ε, ασφάλεια των τροφίμων και την προέλευση των προϊόντων και θα συμφωνήσω με αυτά που είπε η τελευταία ομιλήτρια. Και θέλω να προσθέσω και το εξή. Η συζήτηση αυτή ε, έχει προκύψει γιατί μας το ζητάνε οι καταναλωτές. Το 70% ζητάει να μας πούνε από πού προέρχονται αυτά τα οποία καταναλώνουν. Και επομένως ε, υπάρχουν και άλλοι λόγοι για τους οποίους πρέπει να υπάρχει αναγραφή. Ε, επίσης, επιμένω ότι έχει σημασία και έχει σχέση με την ασφάλεια των τροφίμων και νομίζω ότι αυτοί οι οποίοι που θεωρούνται ότι είναι η πιο ποιοτική παραγωγή είναι αυτοί που έχουν τις περισσότερες δυνατές πληροφορίες. Και πρέπει να φτάνουν σε όλους γιατί αλλιώς θα υπάρχει θέμα ανισότητας. Θεωρώ ότι είναι καλή λοιπόν ε, η ευκαιρία αυτή να συζητήσουμε το θέμα αυτό και την ανάγκη να υπάρχουν περισσότερες πληροφορίες όσο το δυνατόν περισσότερο στην ετικέτα, όχι μόνο για τα τρόφιμα, για όλα τα τρόφιμα, είτε οι προέρχονται από την Ευρωπαϊκή Ένωση είτε εκτός. Ευχαριστώ. Η κυρία Σούισα. grupe Λοιπόν, παρακολουθώ τη συζήτηση και διαπιστώνω πως όλοι εμείς που εκπροσωπούμε του Ευρωπαίου πολίτε έχουμε, αν και έχουμε τον κοινό στόχο να του εκπροσωπήσουμε, έχουμε διαφορετικέ αντιλήψεις και διαφορετικέ προσεγγίσει. Οι διάφορε μελέτε που έχουμε στα χέρια μα καταλήγουν σε διαφορετικά συμπεράσματα, διαφέρουν πολύ μεταξύ του. Γι' αυτό δυσκολεύομαι να τι εμπιστευτώ. Και θα ήθελα ε, η Επιτροπή να διεξάγει εκείνη μια δική της έρευνα για να γνωρίζουμε ακριβώς πόσο θα επηρεαστεί η τιμή του προϊόντος από το να γίνει υποχρεωτική η αναγραφή. Γνωρίζουμε από το Ευρωβαρόμετρο, από άλλες μελέτες, ότι οι Ευρωπαίοι ε, καταναλωτές επιθυμούν να γνωρίζουν την προέλευση. Αλλά αυτό δεν απαντάει στο ερώτημα εάν ε, η αναγραφή πρέπει να είναι υποχρεωτική ή προαιρετική. Γι' αυτό ζητώ από την Επιτροπή να διεξάγει εκείνη ακόμα μια έρευνα που να μας απαντήσει ακριβώς τι επιθυμούν οι Ευρωπαίοι πολίτες. Γιατί δεν θέλω να λάβουμε μια απόφαση απλώς επί τη βάση των πολιτικών μας ιδεολογιών, αλλά επί τη βάση των επιθυμιών των Ευρωπαίων πολιτών. Πρέπει να καταλάβουμε ακριβώς τι επιθυμούν και να τους ε, υπηρετήσουμε. Νομίζω το ζήτημα εδώ δεν είναι απλώς η διαφάνεια. Υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ των προϊόντων από τις ανατολικές χώρες και από τις δυτικές χώρες. Και αυτό είναι ένα ζήτημα το οποίο δεν μπορούμε να το αποκρύπτουμε, καλύτερα να το συζητήσουμε. Πάντως δεν έχουμε αρκετά στοιχεία στη διάθεσή μας, πιστεύω, για να το συζητήσουμε το θέμα και ζητώ από την Επιτροπή να μας τα παράσχει κάποια στιγμή. Ο κύριος Εκ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, η προαιρετική αναγραφή δεν βοηθάει τον καταναλωτή. Λέμε ότι καλή εμπιστοσύνη αλλά καλύτερος ο έλεγχος. Έχουμε δει στο παρελθόν πόσα σκάνδαλα υπήρξαν στον τομέα των τροφίμων. Όταν χρησιμοποιούνται γαλακτοκομικά και κρέα σε μεταποιημένα τρόφιμα θα πρέπει ε, να αναφέρεται η χώρα καταγωγή. Έχουν δικαίωμα στι πληροφορίε αυτέ οι καταναλωτέ, και είναι υποχρέωση της Κομισιόν ε, να αντιμετωπίσει την απάτη στον τομέα των τροφίμων. και πιστεύω ότι το κόστος που υπολογίζεται είναι υπερβολικό. Υπάρχουν υπολογισμοί από ε, την Γερμανία, από την εταιρεία Φρόστερ, που δείχνει ότι μπορεί να γίνει με οικονομικό τρόπο η αναγραφή της χώρας καταγωγής. Έρευνα του 2013 δείχνει ότι το 30% των ε, ερωτηθέντων βρίσκουν ότι είναι πολύ ε, σημαντικό να αναγράφεται η χώρα καταγωγής. Ε, η επισήμαση αυτή τη στιγμή δεν ε, ανταποκρίνεται στις επιθυμίες των καταναλωτών. Είναι πολύ καλύτερο να ενημερώνεται ο καταναλωτής και μόνος τον αποφασίζει εάν θέλει τοπικά, εγχώρια ή εισαγόμενα προϊόντα. Και μία ακόμα παρατήρηση που έκανε και μία συνάδελφος εδώ μπροστά. Η υποχρεωτική αναγραφή είναι και προώθηση των τοπικών προϊόντων. Τα τοπικά προϊόντα σημαίνουν λιγότερος χρόνος μεταφοράς ε, των ζώων ε, και των προϊόντων, άρα λιγότερο κόστος. Υπάρχουν ε, λοιπόν ε, πολύ βάσιμα επιχειρήματα για την υποχρεωτική αναγραφή. Η Κομισιόν θα πρέπει να ακούσει περισσότερο τους καταναλωτές και λιγότερο τις επιθυμίες της βιομηχανίας τροφίμων. Η κυρία Εράντς Κυρία Εράντς, ευχαριστώ. Εγώ νομίζω ότι στο θέμα αυτό πρέπει λίγο να πριτανεύσει η λογική. Είστε mejor? Καλύτερα με αυτό. Εντάξει. Έλεγα λοιπόν ότι στο θέμα αυτό θεωρούμε ότι πρέπει να πριτανεύσει η λογική και να υπάρχει μια ισορροπία. Συγγνώμη, έχασα και τα χαρτιά μου. Πρέπει λοιπόν να δούμε τι επιθυμούμε και τι μπορούμε να υλοποιήσουμε. Αφενός πρέπει να γνωρίζουμε ότι ένα προϊόν Εάν πραγματικά θέλουμε να γνωρίζουμε την προέλευση ενός προϊόντων, μάλλον να το πω αλλιώς, γιατί θέλουμε να κάνουμε διάκριση μεταξύ ενός ελαφρώς μεταποιημένου προϊόν και ενός πραγματικά μεταποιημένου προϊόντος. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ένα φρέσκο λουκάνικο ε, πρέπει να συμπεριλαμβάνεται σε αυτό τον κατάλογο και όχι ένα λουκάνικο Φραγκφούρτης, αν πραγματικά θέλουμε να ξέρουμε όλη την προέλευση όλων των προϊόντων. Επίσης, θεωρώ ότι είναι πολύ λογικό να μην υπάρχουν όρια, γιατί ε, η χώρα είναι το όριο ε, που θέτουμε. Γιατί να μην λέμε από ποιο χωριό ή από ποια περιοχή είναι ένα προϊόν. Μας ξεφεύγει λίγο η κατάσταση από τα χέρια νομίζω. Όταν έχουμε ένα προϊόν με ε, ε, προστατευόμενη ονομασία προέλευσης, είναι pop ή γεωγραφική ένδειξη, τότε γνωρίζουμε από πού προέρχεται ένα προϊόν. Ένα προϊόν προστατευόμενης ονομασίας προέλευσης ε, πρέπει να περιλαμβάνει συστατικά που προέρχονται από την περιοχή που προβλέπει η γεωγραφική ένδειξη. Αλλά το να τα πάμε παραπέρα για τα προϊόντα για μένα είναι τρέλα και θεωρώ ότι το όριο θα πρέπει να είναι να υπάρχει μια προστιθέμενη αξία για τις προσπάθειες που ήδη κάνουν ε, οι παραγωγοί. Θα μπορούσαμε ίσως να μιλάμε για προϊόντα εντός ή εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κατ' εμέ αυτό είναι το ανώτατο όριο. Γιατί το άλλο πραγματικά μου φαίνεται ότι υπερβαίνει τα όρια και απαιτούμε πολύ μεγάλη προσπάθεια, διότι το είπαν και κάποιοι από τους συναδέλφους, κάποιος ο οποίος παράγει ε, πρώτη ύλη ε, και χρησιμοποιεί από εκεί και πέρα προϊόντα για μεταποίηση. Το να γνωρίζουμε την πρώτη ύλη ε, όλος, όλων των προϊόντων είναι πάρα πολύ δαπανερό. Πρέπει να αλλάζει ετικέτα, πρέπει να αλλάζουν διαδικασίες, πρέπει να αλλάζει τεκμηρίωση. Δεν είναι τόσο εύκολο, δεν βάζουμε απλώς μια ονομασία σε μια ετικέτα και τελείωση. Είναι πολλά περισσότερα πράγματα. Ε, τι θα αλλάξει για μένα εάν ένα προϊόν από το Πακιστάν ή από το Εκουαντόρ. Θέλω απλώ να είναι βάση προδιαγραφών. Δεν με ενδιαφέρει τόσο πολύ από το που προέρχεται. Τι σημασία έχει αν είναι ένα περολάχιστο τμήμα ενό μεταποιημένου προϊόντο. Ε, το, για μένα θα έπρεπε να είναι εντό ή εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση η διάκριση. Και όποιο θέλει να το κάνει και θέλει πραγματικά να μα λέει στην ετικέτα του τι, από πού είναι ένα προϊόν, μπορεί να το κάνει. Είναι προαιρετικό και επιτρέπεται. Ε, Έχουμε τους παραγωγούς και αυτούς που αγοράζουν τα προϊόντα. Και πρέπει να σας πω ότι αυτό το οποίο έχει σημασία για θέματα ασφαλείας έχει ήδη ρυθμιστεί. Ε, υπάρχει υποχρέωση για παράδειγμα ε, να ξέρουμε πού ανατράφηκαν και πού υπήρξε η σφαγή των ζώων γιατί ήταν σημαντικό για την ε, ε, ε για τη διατροφική ασφάλεια για την ασφάλεια των τροφίμων συγγνώμη. Και μέχρι εκεί μπορούμε να πάμε, γιατί αν πάμε παραπέρα είναι σαν να θέλουμε όρια στην παραγωγή των προϊόντων και δεν νομίζω ότι οι καταναλωτές είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν για αυτά τα όρια. Ευχαριστώ. Η κυρία Σεγκέρ Σας ευχαριστώ. Έχω ακούσει όλους τους ε, συναδέλφους και τα επιχειρήματα και κυρίως το επιχείρημα της τιμής, αλλά δεν είναι αυτό το πιο σημαντικό. Το ζήτημα είναι το, ε, για εμένα το πιο σημαντικό είναι το ζήτημα του ελέγχου. Ποιος θα ελέγξει πραγματικά ότι η προέλευση είναι όντως αυτή που αναγράφεται. Γιατί δεν πρόκειται μόνο για μια περιορισμένη αγορά, πρόκειται για μια αγορά η οποία όλο και αυξάνει. Η αγορά δηλαδή των ε, ποιοτικών τροφίμων. Θα πρέπει λοιπόν να λάβουμε υπόψη μας και τις δυσκολίες που θα δημιουργήσει η εισαγωγή μια τέτοιας διαδικασίας ελέγχου και τελικά κατά πόσο ο καταναλωτής θα είναι διατεθειμένος να πληρώσει την ε, αυξημένη τιμή που θα, ε, στην οποία θα οδηγηθούμε εξαιτία αυτής της διαδικασίας. Υπάρχουν παραδείγματα από ε, χώρες στις οποίες εφαρμόστηκε αυτό και σε ορισμένους τομείς. Δεν γνωρίζω όμως πώς θα μπορούσαμε να προχωρήσουμε. Ο Πρόεδρος. Τώρα θα δώσω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στην κυρία Γιούλκα. Σας ευχαριστώ. Και σας ευχαριστώ επίσης για αυτή την ε, ενδιαφέρουσα και ζωντανή συζήτηση. Θα ήθελα απλώς να υπενθυμίσω τα εξής. Ο κανονισμός για την υποχρεωτική ε, ετικετοθεσία έχει ήδη επεκταθεί και εφαρμόζεται πλέον και σε νέες κατηγορίες τροφίμων, δηλαδή πέρα από το μοσχαρίσιο κρέας, τώρα πλέον ε, συμπεριλαμβάνονται και τα εγωπρόβατα και το χοιρινό και το, ε, και το κοτόπουλο. Μια σημαντική λοιπόν επέκταση αυτού του κανονισμού Επίσης η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έκανε μια μελέτη ε, που εξέταζε το κατά πόσον θα, είχε, θα ήταν σκόπιμο να γίνει υποχρεωτική η αναγραφή για τα γαλακτοκομικά, τα προϊόντα του γάλακτος και τα προϊόντα του κρέατος και κατ' ουσία το συμπέρασμα ήταν ότι η καλύτερη επιλογή είναι η προαιρετική αεθελοντική αναγραφή γιατί αυτή δίνει τη δυνατότητα στους καταναλωτές, εάν το επιθυμούν, να επιλέγουν τρόφιμο από μια συγκεκριμένη γεωγραφική προέλευση, χωρίς όμως να ε, επιβάλλει ε, το κόστος και την πολυπλοκότητα της διαδικασίας σε όλους τους παραγωγούς και σε όλες τις ε, εταιρείες που δραστηριοποιούνται στον κλάδο των τροφίμων. Θα έλεγα ότι δεδομένης και της οικονομικής κατάστασης ε, δεν θα πρέπει να υποβαθμίζουμε το ζήτημα του κόστους. Θα πρέπει να το θυμόμαστε. Επίσης, υπενθυμίζεται ότι το μερίδιο της αγοράς των τροφίμων που φέρουν σήμανση προέλευσης είναι μικρό. Το οποίο δείχνει ότι οι καταναλωτές δεν είναι διαταθειμένοι ε, να πληρώσουν το αυξημένο κόστος που θα είχε μια γενικευμένη αναγραφή. Συζητήθηκε λοιπόν το ζήτημα του κόστους ε, και για τους καταναλωτές και για τους, τις ε, εταιρείες. Τα στοιχεία ε, αντιφάσκουν. Και βεβαίως θα πρέπει να μην δεχόμαστε χωρίς να τα επεξεργαζόμαστε τα στοιχεία που μας δείχνει η ίδια η, ίδια η βιομηχανία των τροφίμων. Βέβαια, γνωρίζουμε ότι, και αυτό δεν αμφισβητείται, ότι θα δημιουργήσει προβλήματα στην ανταγωνιστικότητα των προϊόντων μας διεθνώς και θα αυξηθεί το κόστος γενικά. Τώρα, όσον αφορά τα μεταποιημένα προϊόντα κρέατος και γαλακτοκομικά, η Επιτροπή θα ήθελε να επισημάνει ότι είναι δύσκολο να καθοριστεί τι ακριβώς σημαίνει ελαφρώς ε, μεταποιημένο τρόφιμο, περισσότερο μεταποιημένο τρόφιμο, θα ήταν δύσκολο να, να δώσουμε τέτοιου τύπου ορισμούς. Επίσης, ας μην ξεχνούμε ότι για ένα μεταποιημένο τρόφιμο, ιδιαίτερα ένα ελαφρώς μεταποιημένο τρόφιμο, ε, η παραγωγή συχνά, μάλλον οι, οι, εταιρείε που το παράγουν συχνά επιλέγουν παραγωγούς από διαφορετικές περιοχές και δεν θα πρέπει να περιορίσουμε αυτή την ευελιξία τους. Θεωρήσε λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι θα πρέπει οποιαδήποτε νομοθεσία στον τομέα αυτό να παραμείνει αναλογική σε κάθε περίπτωση όταν υπάρχει ε, αναγραφή ε, αυτή δεν πρέπει να είναι παραπλανητική και έχουμε ήδη αντιμετωπίσει ζητήματα παραπλάνησης των καταναλωτών, θα επανέλθω σε αυτό. Προκρίνουμε λοιπόν τη, τη λύση της ενθελοντικής αναγραφής της προέλευσης όταν Επίσης υπάρχει η περίπτωση όπου το κύριο συστατικό είναι διαφορετικό, έχει διαφορετική προέλευση από την προέλευση των υπολείπων συστατικών, αυτό θα πρέπει να αναγράφεται. Η Κομισιόν θα επανεξετάσει ε, αυτούς τους, ε, τους κανόνες εν χρόνο, ε, τους κανόνες δηλαδή για την εθελοντική αναγραφή. Θέλω επίσης να σταθώ σε δύο άλλα σημεία. Πρώτον το ζήτημα της ασφάλειας των τροφίμων που αναφέρεται. Η Επιτροπή θεωρεί ότι η ασφάλεια των τροφίμων θα πρέπει να γίνεται ε, σεβαστή και θα πρέπει να ε, την εξασφαλίζουμε ανεξαρτήτως του εάν θα αναγράφεται η προέλευση, επομένως δεν συνδέονται αυτά τα δύο ζητήματα. Επίσης, είναι άλλο το ζήτημα όταν υπάρχει απάτη, μιας και αναφέρθηκε και το πρόβλημα με το κρέας αλόγου. Και επισημαίνουμε ότι ακόμα και αν υπήρχε υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης, το σκάνδαλο με το κρέας αλόγου δεν θα είχε αποφευχθεί. Ήταν άλλη τάξεως ε, η απάτη σε αυτήν την περίπτωση. Δηλαδή η υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης ενός προϊόντος δεν θα εξαλείψει τις απάτες. Το ζήτημα και ο μόνος τρόπος αντιμετώπισης αυτών των πρακτικών είναι να υπάρχουν σωστοί επίσημοι έλεγχοι από τους φορείς ελέγχου τροφίμων. Κάτι ακόμα. Η χνηλασιμότητα σε όλη την διατροφική αλυσίδα. Αυτό είναι υποχρεωτικό, είναι δεδομένο η χνηλασιμότητα είναι ένας από τους κυριότερους στόχους που ε, απαιτείται να ε, τηρεί ε, η βιομηχανία των τροφίμων. Είναι εφικτή η χνηλασιμότητα και διασφαλίζεται, αλλά αυτό δεν οδηγεί κατά σε υποχρεωτική αναγραφή της προέλευσης των διαφόρων συστατικών στις ετικέτες που φτάνουν στον καταναλωτή. Σας ευχαριστώ. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστώ να σας υπενθυμίσω την προθεσμία των τροπολογιών στο ψήφισμα. 12 η ώρα 1η ε, Μαρτίου. Στην Επιτροπή θα έρθει στις 22 ε, ε, Μαρτίου και 2 Απριλίου στην Ολομέλεια. Και προχωράμε στο επόμενο θέμα της ημερήσιας διάταξης, εφαρμογή της νομοθεσίας σχετικά με την υγεία. Ως συνήθως, θα δώσουμε πρώτα το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει στα ερωτήματα τρία λεπτά αναερώτηση ή λιγότερο αν είναι δυνατόν, διότι πάντα μας πιέζει ο χρόνος. Και κατόπιν ε, θα δώσουμε το λόγο στον βουλευτή που έχει θέσει την ερώτηση. Γενική Διεύθυνση Σαντέ, ο κύριος παρακαλώ, για την πρώτη ερώτηση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε να κάνω πρώτα κάποιες γενικές παρατηρήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 4 Σεπτεμβρίου του περσινού έτους ε, ε, εξέδωσε την έκθεση σχετικά με την εφαρμογή της ε, οδηγίας. Καλύπτονται οι πιο βασικές διατάξεις όπως είναι η κινητικότητα των ασθενών, η επιστροφή των δαπανών κλπ. Η επόμενη έκθεση έχει προγραμματιστεί για το 2018. Η έκθεση συζητήθηκε ήδη κατά την ανεπίσημη υπουργική, άτυπη υπουργική συνεδρίαση στο Λουξεμβούργο. Τι έχουμε κάνει λοιπόν ε, κατά την ε, εκπόνηση της έκθεσης αυτής. Καταρχάς, πήγαμε στις πρωτεύουσες όλων των κρατών μελών, ε, συζητήσαμε σε τεχνικό επίπεδο διάφορα θέματα που σχετίζονται με την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Είχαμε συναντήσεις και με διάφορους ενδιαφερομένους σε κάθε πρωτεύουσα. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί με τα κράτη-μέλη ότι η συλλογή δεδομένων για την κινητικότητα των ασθενών, για την προηγούμενη έγκριση κλπ. Ε, είναι πολύ σημαντική επίσης. και όσον αφορά την ε, συλλογή πληροφοριών σχετικά με τα εθνικά σημεία επαφής. 26 από 28 κράτη-μέλη υπέβαλαν τέτοια δεδομένα. Εξετάζονται οι καλές πρακτικές ε, και τα πιθανά εμπόδια για την διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Εξετάζονται επίση ε, τα δικαιώματα των ε, ασθενών, τα πρότυπα που εφαρμόζονται στα άλλα κράτη-μέλη, η διαδικασία για την επιστροφή δαπανών, η ύπαρξη ε, αξιόπιστων πηγών δεδομένων, καθώς και την επιλογή των, καλύτερων, των χωρών με τις καλύτερες συνθήκες. Το 2014 είχαμε έρευνα του ε, Ευρωβαρόμετρου σε συνέχεια μιας παρόμοιας ε, έρευνας που είχε γίνει το 2007. Υπάρχει ευαισθητοποίηση σχετικά με το δικαίωμα των ε, μάλλον η ευαισθητοποίηση των ασθενών σχετικά με τις δυνατότητες υγειονομικής περίθαλψης σε άλλη χώρα παραμένει χαμηλή. Δύο στους δέκα γνωρίζουν τα δικαιώματα αυτά και μόνο ένας στους δέκα γνωρίζει ποιο είναι το εθνικό σημείο επαφής παρότι υπάρχουν διακυμάνσεις από χώρα σε χώρα. Η έρευνα σχετικά με τον πειραματικό σχεδιασμό ε, ανατέθηκε το 2014 και δημοσιεύθηκε το 2015 και εξετάζει τις επιλογές των ασθενών με βάση την ε, οδηγία. Προσπαθούσε η έρευνα να εξετάσει ποιοι παράγοντες επηρεάζουν ε, τις επιλογές των ασθενών κατά την ε, επιλογή διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Ε, ε, φυσικά τα στοιχεία αυτά είναι διαθέσιμα. Από τον Δεκέμβριο του 2013 μέχρι τον Ιανουάριο 2014 είχαμε σχετικές διασκέψεις στις Βρυξέλλες, Λιουμπλιάνα, Αθήνα και Ταλίν. Και τέλος, όσον αφορά την μεταφορά της ε, οδηγίας ε, στο εθνικό δίκαιο, εξετάστηκε η κατάσταση σε 20 κρατη Αυτά λοιπόν έγιναν σε προετοιμασία της έκθεσης αυτής. Ε, να σας πω και λίγα λόγια σχετικά με τη μεταφορά στο εθνικό δίκαιο της οδηγίας. Η Κομισιόν εξετάζει σε τι βαθμό έχει ε, εφαρμοστεί η οδηγία. Κατά 26 κρατών μελών ξεκίνησαν διαδικασίες ε, παράβασης λόγω ε, λοιπούς εφαρμογής. Αυτή τη στιγμή έχει εφαρμοστεί σχεδόν πλήρω η οδηγία σε όλα τα κράτη-μέλη τη Ευρωπαϊκής Ένωσης. Για παράδειγμα υπάρχουν σημεία επαφή σε όλα τα κράτη-μέλη που παρέχουν πληροφορίε προ του ασθενεί για θέματα ποιότητα και ασφάλεια. Επίση, όλα τα κράτη-μέλη συμμετέχουν στον ε, μηχανισμό συντονισμού και ε, στο e-health, ε, την ηλεκτρονική υγεία. πιο δύσκολο είναι το να διαπιστώσουμε πώς έχει εφαρμοστεί η οδηγία λόγω της διαφοράς ανάμεσα στα διάφορα εθνικά συστήματα σε εθνικό επίπεδο διαπιστώσαμε ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες για κάποια κράτη-μέλη. Για παράδειγμα, υπάρχουν πολύπλοκα συστήματα προηγούμενης έγκρισης που μπορούν να αποτελέσουν εμπόδιο για ασθενείς από άλλε χώρε. Ή ε, χαμηλά, ε, ε, χαμηλό ποσοστό επιστροφής των δαπανών. Το Ευρωπαρόμετρο δείχνει ότι Ε, οι Ευρωπαίοι πολίτες ε, συνεχίζουν να μην γνωρίζουν πολλά σχετικά με τις δυνατότητες ε, διασυνοριακής υγειονομικής περίθαλψης. Γι' αυτό η πρόκληση για μας είναι να φροντίσουμε για την περαιτέρω εφαρμογή της οδηγίας. Σας διαβεβαιώ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα λάβει υπόψη της τα ευρήματα αυτά στην επόμενη φάση. Σας ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γκροστέτ είχε θέσει την ερώτηση. Θέλετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η ερώτησή μου έχει να κάνει με το Ευρωπαϊκό ε, Δίκτυο Κέντρων Αναφοράς, διότι στην επόμενη πρόσκληση υποψηφιότητας ε, για τα κέντρα αναφορών θα γίνει εντός του έτους ε, και θα ήθελα να ξέρω τι μπορεί να κάνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να βελτιώσει την ενημέρωση για το Ευρωπαϊκό Δίκτυο και να ενθαρρύνει τη συμμετοχή των καλύτερων κέντρων αριστείας. Μεταξύ άλλων την Ευρωπαϊκή Επιτροπή Εμπειρογνωμόνων Σπανίων Ασθενών που ε, γνωμοδότησε το 2011 για την δημιουργία ενός κέντρου εμπειρογνωμοσύνη όσον αφορά τις σπάνιες ασθένειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και θα ήθελα να ξέρω πού βρισκόμαστε στην εφαρμογή αυτής της σύστασης. Ε, αυτά από πλευράς μου. Να σας πω επίσης ότι θα πάρω και το λόγο ε, εξ ονόματος του κυρίου Πέτερλε που είχε κάποιες ερωτήσεις ε, όταν θα φτάσουμε στο θέμα και αν θέλετε να μου ξαναδώσετε το λόγο. Ωραία, η κυρία Σαϊαρπέδη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προσθέτω ερώτηση εξ ονόματος της Μέρη Μαγκίνες. Ε, σύμφωνα με την έρευνα του Ευρωβαρομέτρου του Μαΐου του 2015, ένα 2% των Ευρωπαίων ε, αναζητούν ε, θεραπεία στο εξωτερικό. Ίσως να μην δίνονται σωστές πληροφορίες σε εθνικό επίπεδο για την διασυνοριακή αναζήτηση κέντρου θεραπείας και θα ήθελα να ξέρω τι γίνεται με τα εθνικά κέντρα επαφής ε, και ε, πώς μπορούμε να ενημερώνουμε καλύτερα τους πολίτες όσον αφορά τα δικαιώματά τους. Αυτή είναι η ερώτηση που θα ήθελα να θέσω. Ευχαριστώ. Voilà, donc, effectivement, euh, je... Ναι, λοιπόν, είναι σημαντικό να είναι ξεκάθαρο πώς θα οργανώσουμε τη συζήτησή μας. Συζητάμε το πρώτο ερώτημα. Ε, εσείς αναφερθήκατε σε ένα θέμα στο οποίο θα, το οποίο θα συζητήσουμε μετά. Υπενθυμίζω λοιπόν ότι η συζήτηση αφορά την πρώτη ε, ερώτηση. Επομένω, θα δώσω το λόγο σε εκείνους που επιθυμούν να τοποθετηθούν επ' αυτής. Η κυρία Ριβαζή, ε, συνεχίζοντας το ερώτημα της κυρίας Γκοστέτς, θέλω να ρωτήσω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή αυτά τα ε, κέντρα, τα ερευνητικά, αναφερθήκατε στο κέντρο για τις σπάνιες ασθένειες. Την προηγούμενη εβδομάδα είχαμε μια συνάντηση για, για ειδικές μορφές θεραπείας όταν κάποιο έχει προσβληθεί από ιό. Αυτή τη στιγμή κάποιο που έχει προσβληθεί από έναν ιό ε, Α, και θέλει να του δώσουμε τη δυνατότητα να θεραπευθεί μέσω ε, ε, ε φαγοβακτηριδίων. Ε, ε, αυτή είναι η μορφή της θεραπείας. Αυτή τη στιγμή πρέπει να πάει στη Γεωργία. Και το ερώτημά μου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είναι τι έχουμε κάνει για να δημιουργηθεί ένα τέτοιο Ευρωπαϊκό Κέντρο Αναφοράς. Αφού έχουμε τη δυνατότητα στη, διάθεσή μας, γιατί δεν έχουμε οργανώσει ακόμα ένα Ευρωπαϊκό Κέντρο ε, Αναφοράς. ευχαριστώ. Κύριε Σφαρία. Το ερώτημα μου και το δικό μου απευθύνεται στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Αναφερθήκατε στην οδηγία για τη διοσυνεριακή περίθαλψη. Προσπαθεί αυτή η οδηγία να προωθήσει και την συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών και την ε, παροχή υψηλής ποιότητας υπηρεσιών υγείας διασυνοριακά. Αναφερθήκατε στα προβλήματα που υπάρχουν στα κράτη-μέλη όσον αφορά την εφαρμογή αυτής της οδηγίας. Στο άρθρο 8 της οδηγίας, 8.5, παράγραφος 5, τονίζεται ότι όταν η υγειονομική περίθαλψη δεν μπορεί εντός εύλογου χρονικού διαστήματος να παρασχεθεί ε, στην επικράτεια του κράτους μέλους και όταν υπάρχει ε, αντικειμενικός ε, λόγος που τεκμηριώνεται ιατρικά με βάση το ιστορικό, τα συμπτώματα, το βαθμό του πόνου στον τον οποίο υφίσταται ο ασθενής και τα λοιπά και τα λοιπά και όλα αυτά αξιολογούνται κατά την υποβολή του ε, αιτήματο. Αναφέρεται λοιπόν στο άρθρο αυτής της οδηγίας ότι θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πόνος που βιώνει ο ασθενής. Το ερώτημά μου είναι, ποια εργαλεία ποιες μεθόδους έχουμε δώσει στα κράτη-μέλη για να μπορέσουν να ανταποκριθούν σε, αυτό το, σε αυτή την απέτηση για να αξιολογούν τον πόνο του ασθενού. Και επίσης γιατί ε, αυτό το ερώτημα που σας θέτω δεν απαντάτε στην έκθεσή σας και αν προτίθεστε να το απαντήσετε σε κάποια μελλοντική έκθεσή σας. Πρόεδρε, ευχαριστούμε τους συναδέλφους. Θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Απαντώ στην κυρία Γκροστέτ και στην ερώτηση της κυρίας Ριβαζή και του κυρίου Φαρία. Τα ευρωπαϊκά δίκτυα αναφοράς είναι ένα από τα πιο σημαντικά εργαλεία συνεργασίας μεταξύ κρατών μελών και τα κλινικά κέντρα αριστείας. Υπάρχουν αρκετά καλά κέντρα σε όλη την Ευρώπη και φυσικά η σωστή ερώτηση είναι πώς θα θέλαμε να συνεργάζονται αυτά. Και η διαδικασία αφενός ε, είναι μια διαδικασία προς τα πάνω αλλά και προς τα κάτω ε, με βάση τους κανονισμούς που τελικώς προτείναμε. Γι' αυτό προσπαθούμε να διασφαλίσουμε ότι αφενός Όσοι ενδιαφέρονται να ε, συστήσουν τέτοια δίκτυα θα πρέπει να είναι ενημερωμένοι και επίση, ε, τα κράτη-μέλη θα πρέπει να γνωρίζουν τι δικαιώματα έχουν για τη συμμετοχή σε αυτή τη διαδικασία. Τώρα, ε, πέρσι όταν καταρτίστηκε αυτό το νέο μοντέλο ευρωπαϊκής συνεργασίας, τι είχαμε κατά νου. Καταρχάς προτείναμε ένα μοντέλο του ευρωπαϊκού δικτύου που είναι ε, κάτι το οποίο προτάθηκε το 2012-2013 και τέθηκε σε δημόσια διαβούληση. Έγιναν ε, αρκετές τεχνικές συνεδριάσεις όπου συζητήσαμε με εμπειρογνώμονες από όλε τις χώρες μέλη για το πώς μπορεί να γίνει αυτή η δουλειά υπήρξαν ε, αρκετές σημαντικές συνεδριάσεις και αναφέρομαι σε δύο συνεδριάσεις ε, πιο συγκεκριμένα. Μία εδώ στις Βρυξέλλες ε, το 2014 και μία στην Πορτογαλία στη Λισαβόνα το 2015. Επομένως είχαμε πάνω από 800 εμπειρογνώμονε κυρίως από τον κλινικό τομέα, αλλά και ενδιαφερόμενους οι οργανώσεις εξειδικευμένες συμμετείχαν σε αυτές τις συνεδριάσεις. Ξεκίνησε μια εξτρεκτή επικοινωνίας η οποία ε, δημοσίευσε αυτή την έννοια των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς και ε, δημοσιεύθηκαν και σε ιατρικά επιστημονικά περιοδικά, σε πάνω από 20 περιοδικά και νομίζω ότι υπάρχει και μια πολύ καλή ιστοσελίδα στην οποία προσπαθούμε να έχουμε και επικοινωνία με τους ενδιαφερομένους και ε, κυρίως διευθυντές κλινικών κέντρων και κράτη-μέλη. Το νομικό πλαίσιο καθορίστηκε το Μάρτιο του 2014 μέσω των πράξεων κατοξουσιοδότηση και εκτελεστικών πράξεων για να δούμε πώς θα λειτουργήσει το σύστημα και τέλος ε, συνεργαζόμαστε στενά με τα κράτη-μέλη και το ε, Διοικητικό Συμβούλιο των Ευρωπαϊκών Δικτύων Αναφοράς, όπου σας είπα ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό και συμμετέχουν όλα τα κράτη-μέλη σε αυτό. Επίσης υπάρχει ένας άλλος σημαντικός φορέας, η Επιτροπή των Σπάνιων Ασθενειών με την οποία προσπαθούμε να εξετάσουμε τις καλύτερες λύσεις και για αυτές τις ομάδες ασθενών. Πώς μπορούμε να οργανώσουμε το σύστημα για αυτούς. Τώρα φτάνουμε σε αυτή τη χρονική συγκυρία στην οποία θα ξεκινήσει η πρόσκληση για υποψηφιότητες. Επομένως ε, έχουμε προετοιμάσει τα πάντα και ελπίζουμε ότι η πρόσκληση θα ανακοινωθεί ε, τη δεύτερη εβδομάδα του Μαρτίου και από εκεί και πέρα θα δούμε πόσο γρήγορα και καλά μπορούν να ε, οργανωθούν αυτά τα δίκτυα. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το γεγονός ότι θα πρέπει να συμμετέχουμε ενεργά με όλους τους διοργανητές αυτών των δικτύων ε, και προσπαθούμε να βοηθήσουμε και σε εθνικό επίπεδο ε, με τους εμπειρογνώμονες και τους εκπροσώπους των κρατών μελών και να συνεργαστούμε και με τα εθνικά κλινικά κέντρα και να προσπαθήσουμε να βοηθήσουμε εκεί. Ελπίζω λοιπόν μέχρι το τέλος του έτου να είμαστε σε θέση να έχουμε τα πρώτα δίκτυα και από εκεί και πέρα οι ασθενείς να είναι σε θέση να ασκήσουν τα δικαιώματά τους ε, με αυτό το νέο πάρα πολύ ευρωπαϊκό σύστημα. Όσον αφορά τώρα τη συγκεκριμένη ερώτηση της κυρίας Ριβαζή, ε, προφανώς ε, και δεν αποφασίζουμε τώρα ποιο κέντρο θα συσταθεί και τι δίκτυο θα συσταθεί. Αυτές είναι ε, για τους ε, διευθυντές, τους διαχειριστές, ε, τα κράτη-μέλη. Αυτοί είναι αυτοί οι οποίοι θα δημιουργήσουν την όλη διαδικασία και θα δούμε τι θα προκύψει και αν από εκεί θα υπάρξουν συγκεκριμένες θεραπείες που θα συμπεριληφθούν σε εξειδικευμένα κέντρα γιατί μπορεί να υπάρχει ένα κέντρο που να είναι εξειδικευμένο σε κάποιο τομέα και θα δούμε αν θα συμπεριληφθούν και αντίστοιχες μορφές θεραπείας όπως η ε, βακτηριοφάγη. Τώρα, η καθυστέρηση και αυτή η πρώτερη έγκριση, πώς λειτουργεί αυτή η διαδικασία. θυμάμαι ότι όταν γίνονταν οι τελευταίε διαπραγματεύσεις εδώ στο Κοινοβούλιο, το ζήτημα αυτό ήταν πάρα πολύ σημαντικό και είπαμε ότι πρέπει να παρακολουθούμε στενά από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό το οποίο μπορούμε να κάνουμε τώρα, ε, συμφωνήσαμε με τα κράτη-μέλη να δίνονται στοιχεία. Ε, στην πρώτη έκθεση δεν είχαμε πάρα πολλέ πληροφορίε, πρώτον ε, διότι όπω εξηγήσαμε το σύστημα καθυστέρησε αρκετά σε πολλά κράτη-μέλη και όταν άρχισαν να χρησιμοποιούνται αυτά ε, ήταν αρκετά αργά. Πρέπει μάλλον να τα δούμε στη δεύτερη έκθεση πόσοι ασθενείς μπόρεσαν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα. Επίσης πρέπει να είναι σαφές ότι υπάρχει και μία ε, φεά ζώνη μεταξύ του κανονισμού αυτού και του κανονισμού περί κοινωνικής προστασίας που επιτρέπει να χρησιμοποιηθεί ένα άλλο σύστημα και είναι οι προϋποθέσεις για τους ε, ασθενείς που είναι καλύτεροι σε αυτό το σύστημα, δεν καλύπτονται ε, κάποια θέματα και καλύπτεται το κόστος ταξιδίου, Επομένως, οι ασθενείς επιλέγουν το καλύτερο σύστημα. Πολλά κράτη-μέλη Ιδίως όσον αφορά την ενημέρωση προς τους ασθενείς, μας λένε ότι ακόμα βρισκόμαστε σε μια φαιά ζώνη, μπορεί να προκύψουν πολλά ερωτηματικά γιατί να χρησιμοποιήσω αυτή την οδηγία όταν μπορώ να χρησιμοποιήσω τον κανονισμό που τον προτιμώ ε, ως ασθενής. Ελπίζουμε όμως ότι στην επόμενη ε, έκθεση θα μπορέσουμε να έχουμε περισσότερα από αυτά τα στοιχεία. Και τώρα όταν θα γίνει και ο έλεγχος ε, της μεταφοράς της οδηγίας, όπως σας είπα θα έχουμε και τις διαδικασίες που θα μας επιτρέψουν να ε, κατανοήσουμε καλύτερα τι γίνεται και τι προβλήματα υπάρχουν και αν επιλήθηκαν. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να προχωρήσουμε τώρα στις επόμενες ερωτήσεις. Νομίζω μπορούμε να συζητήσουμε μαζί τα σημεία 2, 3 και 4, διότι σχετίζονται μεταξύ τους. Καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να απαντήσει. Και κατόπιν θα δώσουμε τη ε, δυνατότητα ε, σε αυτούς που υπέβαλαν την ερώτηση να απαντήσουν. Παρακαλώ. I just went through, Οι ερωτήσεις αυτές σχετίζονται με τα εθνικά σημεία επαφής. Και όπως ήδη είπα, είναι πολύ χαμηλό το επίπεδο πληροφόρησης. Και γι' αυτό ως Ευρωπαϊκή Επιτροπή αποφασίσαμε να συνεργαστούμε στενά με τους σχετικούς οργανισμούς. Θα ξεκινήσω από την ερώτηση του κυρίου Πέτερλε σχετικά με την εναρμόνιση των εθνικών σημείων επαφής. Η απλή απάντηση είναι ότι δεν μπορεί να γίνει εναρμόνιση, διότι είναι τόσο διαφορετικές οι χώρες μεταξύ τους. Για παράδειγμα, στο Ηνωμένο Βασίλειο έχουμε τέσσερα διαφορετικά εθνικά σημεία επαφής. Σε κάποιες χώρες υπάρχει ένα. Σε άλλες πρόκειται για μια ομάδα φορέων. Υπάρχουν λοιπόν σημαντικές διαφορές. Προσπαθούμε να διασφαλίσουμε την ανταλλαγή πληροφοριών ώστε να μπορεί να γίνει η ανταλλαγή ιδεών σχετικά με τον βέλτιστο τρόπο λειτουργίας. Γνωρίζω τους ανθρώπους που εργάζονται στους οργανισμούς αυτούς. Είναι πολύ ικανοί και στις 2 Δεκεμβρίου είχαμε τη δυνατότητα συζήτησης ε, του συστήματος συνεργασίας. Δηλαδή πώς, μπορεί, πώς μπορούν να ανταλλάσσονται ερωτήσεις, πώς μπορεί κανείς να ακολουθεί το ιστορικό ενός ασθενούς και πώς μπορεί να αυξηθεί η συνεργασία μεταξύ τους. Προσπαθήσαμε λοιπόν να δούμε πώς λειτουργούν, πώς εργάζονται. Και αναπτύξαμε ένα πρόγραμμα. Είχαμε δίθεν ασθενεί που ζητούσαν πληροφορίες, έπαιρναν τηλέφωνα. Για να δούμε πώς λειτουργούν τα σημεία επαφής. Μπορεί να σας εκπλήσει ότι κάποια από τα κέντρα αυτά δεν χρησιμοποιούν τηλέφωνα. Και βέβαια θα ήταν πάρα πολύ ωραίο να υποβάλλονται όλες οι ερωτήσεις ηλεκτρονικά, αλλά δεν έχουν ε, όλοι πρόσβαση σε email στην Ευρώπη. Αυτό απλά είναι ένα παράδειγμα. Συζητήσαμε και τη χρήση των κοινωνικών μέσων δικτύωσης. Θεωρήθηκε ότι δεν είναι το κατάλληλο μέσο για να δίνονται ατομικές απαντήσεις σε ατομικά προβλήματα. Συχνά χρειάζεται εις βάθος γνώση του προβλήματος τους, του συστήματος ε, στο οποίο βρίσκονται κλπ. Ο κύριος Μπετισίνη έθεσε ερώτηση σχετικά με το επίπεδο επικοινωνίας με διάφορους, επικοινωμένους, ε, με διάφορους ενδιαφερομένους. Συγγνώμη. Υπάρχει οδηγία του Μαρτίου του 2014 που θεσπίζει ότι πρέπει να υπάρχει επικοινωνία με τις ασφαλιστικές εταιρείες Το βασικό ερώτημα είναι μπορούμε να αυξήσουμε την ευαισθητοποίηση όχι μόνο μεταξύ των ασθενών αλλά και μεταξύ των παρόχων υπηρεσιών υγείας και μεταξύ όλων των ενδιαφερομένων φορέων. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στους ε, συγγυρές ξεκινώντας από τη κυρία Κροστέτ. Εδώ εκπροσωπώ τον συνάδελφό μου, τον Τερλέκιν, που δεν μπόρεσε να είναι εδώ απόψε. Είπατε ότι δεν είναι εφικτό να υπάρξει εναρμόνιση των εθνικών ε, σημείων επαφής και μας διαβεβαιώσατε ότι υπάρχει ανταλλαγή πληροφοριών, αλλά ναι, το ζήτημα που τίθεται είναι ποια είναι η ποιότητα των πληροφοριών που δίνονται στους ασθενείς από τα 28 διαφορετικά κράτη-μέλη. Το σημαντικό είναι να επιτύχουμε τον στόχο μας. Δεδομένου λοιπόν ότι δεν μπορεί να υπάρξει εναρμόνιση πλήρης εξαιτία των διαφορών μεταξύ κρατών μελών, πρέπει να εξασφαλίσουμε ότι η, ποιότητα των πληροφοριών που δίνουν και τα 28 κράτη-μέλη είναι εξίσου υψηλή. Θα ήθελα να μου πείτε τι έχετε κάνει προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Εμείς ευχαριστούμε. Μήπως ο κύριος Πετιτσίνη θέλει να προσθέσει κάτι. Ναι, εγώ θέλω να προσθέσω κάτι μικρό. Δεν κατάλαβα πολύ καλά την απάντησή σας, για να είμαι ειλικρινής. Κατάλαβα ότι υπάρχει ένα εθνικό σημείο επαφή στην Ιταλία. Επαληθεύσατε όμως εσείς από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής ότι λειτουργεί γιατί για μας ε, δεν υπάρχει κανένα ενεργό κέντρο για τους πολίτες, δεν υπάρχει αριθμός τηλεφώνου, ιστοσελίδα, ε, αριθμός διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου για τους πολίτες. Επίσης ε, δεν συμμετείχαν οι πολίτες και οι ασθενείς για την δημιουργία του σημείου επαφής που είναι κάτι το οποίο αναφέρεται ρητός στην οδηγία. Ευχαριστώ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν επιπλέον ερωτήσεις από τους πολύπους. Ωραία. Μπορούμε να δώσουμε πάλι το λόγο στην Επιτροπή για να απαντήσει. Θα ξεκινήσω από την απάντηση προς τον κύριο Πεντιτσίνη. Ναι, η Ιταλία έχει συμπεριληφθεί σε αυτή τη διαδικασία ψευδοασθενών όταν ε, ψευδοασθενείς ε, καλούσαν σε διάφορα ε, κέντρα και κάναμε μια τυχαία ε, επιλογή και υπάρχει απάντηση. Δεν δημοσιεύουμε στοιχεία χώρα... αλλά η Ιταλία είναι ενήμερη για το τι ακριβώς συμβαίνει. Όπως σας είπα δεν υπάρχει πρόσβαση μέσω τηλεφώνου στην Ιταλία και το θέσαμε το ζήτημα αυτό, αλλά γιατί δεν είναι μόνο η Ιταλία αλλά και κάποια άλλες χώρες μέλη δεν ε, προσφέρουν δυνατότητα πρόσβασης μέσω τηλεφώνου. Είμαστε σε επαφή μαζί τους, τους ξέρουμε, υπάρχουν, ε, μην νομίζετε. Επιτρέψτε μου λοιπόν να σας απαντήσω αυτό. Τώρα, όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας Γκροστέτ, αυτό είναι το θέμα, όντως, τι κάνουμε. Ε, διασταυρώνουμε τους ελέγχους μας ε, σε αυτή τη διαδικασία, προσπαθούμε να δούμε ε, παραδείγματα από διάφορα εθνικά σημεία επαφής. Ε, να σας παραπέμψω στην παρουσίαση της Γερμανίας όταν τέθηκε θέμα του πώς ενημερώνεις για την ποιότητα των ε, ε, ιδρυμάτων και την ασφάλεια των ασθενών. Είναι πολύ καλά ανεπτυγμένο το σύστημα εκεί. Και επίσης τίθεται και το θέμα της πόση εμπειρία διαθέτει κάποιος, τι πρόσβαση σε γνώσεις υπάρχει από αυτούς που παρέχουν υπηρεσίες υγείας. Και στην ουσία πόσα μπορείς να επενδύσεις στην ανάπτυξη αυτών των μοντέλων. Φυσικά έχει σημασία να γίνουν επενδύσεις, διότι ο αριθμός των ασθενών που αναζητούν ε, ε, μια θεραπεία μπορεί να αυξηθεί και επίσης επειδή σε κάποιες χώρες εξήγησαν ότι τα εθνικά σημεία επαφής είναι η τελευταία ευκαιρία ε, όταν φτάσουμε στην τελευταία ίστατη λύση, μπορεί οι ε, ασθενείς να λάβουν καλή θεραπεία στη χώρα τους. Ε, παραδείγματος χάρη, ε, χρησιμοποιείται το σύστημα στους συνηγόρους των ασθενών γιατί μπορούν να τους προσφέρουν κάποιες καλές λύσεις. Ε, θέλουν ε, λοιπόν τα κράτη-μέλη να έχουν κατάλληλες λύσεις και τα δημιουργούμε τα συστήματα. Αυτά τα κέντρα, να ξέρετε, τα σημεία επαφή είναι πολύ καινούργια ακόμα και πρέπει σιγά-σιγά να βρουν το βηματισμό τους ε, και να δουν πώς θα λειτουργεί ε, με τον καλύτερο τρόπο. Επίσης βοηθάμε μια τελευταία παρατήρηση με πρόσβαση στο λεγόμενο σύστημα IMI, το σύστημα της εσωτερικής αγοράς, το οποίο επιτρέπει ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών μεταξύ εθνικών σημείων επαφής. Παραδείγματος χάρη όταν γίνεται γίνεται μια ε, ανταλλαγή πληροφοριών για κάποιον ασθενή μπορούν να χρησιμοποιήσουν το σύστημα και να ε, γίνει ε, με ασφάλεια ανταλλαγή δεδομένων και φυσικά να υπάρχει και πρόσβαση σε ένα εξειδικευμένο κέντρο. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να περάσουμε στην επόμενη ερώτηση. Εξειδικευμένη φροντίδα. Είναι η πέμπτη ερώτηση. Ο λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Yeah, so, uh, Μάλιστα. Και αυτό ήταν ένα από τα σημαντικότατα ε, στοιχεία στη συζήτηση κατά τη διαπραγμάτευση της οδηγίας. δεν έχουμε και δεν σκοπεύουμε να εκδώσουμε κατευθυντηρίες οδηγίε προς τα κράτη-μέλη. Ανταυτού, αποφασίσαμε να διεξάγουμε μια μελέτη βιβλιογραφική ε, που αφορά στη, στο υψηλού κόστους εξειδικευμένο ιατρικό εξοπλισμό και υποδομές φροντίδας. Η μελέτη αυτή θα δημοσιευθεί ε, στα τέλη Μαΐου φέτος. Και ελπίζω ότι αυτή η μελέτη θα απαντήσει στο ερώτημά σας για το πώς ακριβώς ορίζουμε, καθορίζουμε τι είναι αυτή η εξειδικευμένη φροντίδα και τι συνιστά εξειδικευμένη φροντίδα και ποιος είναι αυτός ο ειδικό εξοπλισμός. Και θα δούμε πώς εφαρμόζουν τα κράτη-μέλη στην πράξη αυτές τις πρόβλεψεις. Ε, υπάρχουν πολλές διαφορετικές μέθοδοι είχε συζητηθεί το ενδεχόμενο να χρησιμοποιήσουμε το οικονομικό κόστος ως στοιχείο που θα μας οδηγήσει στο να ορίζουμε τι είναι εξειδικευμένη φροντίδα, δηλαδή να είναι φροντίδα που κοστίζει πάνω από ένα συγκεκριμένο ποσό, περισσότερο από ένα συγκεκριμένο ποσό, αλλά αποφασίσαμε καλύτερα ε, να ε, ε, δοθεί η δυνατότητα στα κράτη-μέλη να αποφασίζουν εκείνα και μέσω της μελέτης θα γράψουν τις διαφορετικές πρακτικές που τα κράτη-μέλη ακολουθούν. Αυτή είναι η απάντησή μας στην πέμπτη ερώτηση. Ο πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία, η κυρία Γκροστέτ. Και εδώ ε, εκπροσωπώ τον συναδελφό μου, αλλά συμφωνώ και πλήρως μαζί του. Είχαμε πολλές συζητήσεις για τις ε, προηγούμενες ειδικέ εγκρίσεις που χρειάζονται όταν, ε, όταν κάποιος ε, ασθενής πρέπει να μεταβεί σε άλλο κράτος για εξειδικευμένη φροντίδα. Και το ερώτημα και αυτό που μας ανησυχούσε είναι τι γίνεται όταν κάποιο κράτος μέλος συστηματικά αρνείται να παραχωρήσει τέτοια εξουσιοδότηση. Αυτό στην πραγματικότητα καταργεί την οδηγία. Αυτό λοιπόν που θα ήθελα να γνωρίζω είναι το εξή. Ε, μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκοπεύει να δώσει στα κράτη-μέλη κατευθυντήριες οδηγίες που θα ξεκαθαρίζουν τι ακριβώς ε, σημαίνει, τι ακριβώς ορίζουμε ως εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα για την οποία χρειάζεται προέγκριση ε, και πώς θα ε, υπάρχει η απαιτούμενη αιτιολόγηση όταν λαμβάνεται η απόφαση αν θα δοθεί ή όχι αυτή η έγκριση. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις για το σημείο αυτό. Η Κομισιόν έχει το λόγο, παρακαλώ. Όπως εξήγησα, το θέμα της ιεράρχησης είναι σημαντικό. Ήταν κάτι που συζητήθηκε αργά τη νύχτα. Συμπεριλαμβάνεται το θέμα αυτό στο σχέδιο συλλογής δεδομένων. και συμπεριλαμβάνει και το κόστος δαπανηρών ε, θεραπείων. Όταν λάβουμε τα σχετικά δεδομένα θα αντιληφθούμε το μέγεθος του προβλήματος. Η κατάσταση διαφέρει από κράτος μέλος σε κράτος μέλος. Το επόμενό μας βήμα θα είναι να βρούμε τον κοινό παρονομαστή. Θα θέλαμε όμως καταρχάς να ολοκληρώσουμε την έρευνα και να δούμε πώς έχει η κατάσταση αυτή τη στιγμή με τις ε, δαπανηρές θεραπείες και κατόπιν να δούμε ποιο θα είναι το επόμενο μας βήμα. Ευχαριστώ. Προχωράμε στο επόμενο θέμα. Ερώτηση υπαριθμών έξι Ευαισθητοποίηση των ασθενών. Ξαναδίνω το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις ενημερωτικές εκστρατείες όπως άλλωστε είπα και κατά την εισαγωγή μου, χρηματοδοτεί την διοργάνωση διασκέψεων, διοργα... Ε, χρηματοδότησε μάλλον τη διοργάνωση διασκέψεων το 2014 και το 2015. οργανώσεις ασθενών ε, αλλά και οι υπάροχοι υγειονομικής περίθαλψης και άλλοι ενδιαφερόμενοι προσκλήθηκαν να συμμετάσχουν σε αυτές τις τέσσερις διασκέψεις σε τέσσερις διαφορετικές χώρες. Επίσης, ε, έχουμε τυπώσει ενημερωτικό έντυπο σε όλες τις γλώσσες της Ευρώπης ε, και παρέχονται πληροφορίες και στην ιστοσελίδα. Στηρίζουμε τις μη κυβερνητικέ οργανώσεις με μια σειρά δραστηριοτήτων εφόσον το επιθυμούν. Συνεχίζουμε τη συνεργασία με τα εθνικά σημεία επαφής, ώστε να μπορούν να εργάζονται πιο αποτελεσματικά. Και τέλος, με chat στο Facebook, προσπαθούμε να ενημερώνουμε κόσμο. Θα βρείτε στην ιστοσελίδα μας τον σχετικό σύνδεσμο. αλλά όπως σας είπα, τα εθνικά σημεία επαφής κάνουν τη δουλειά τους και εμείς δεν θέλουμε να ξεπεράσουμε τα δικά μας όρια. Thank Σας ευχαριστώ πολύ. Ξαναδίνω το λόγο στην κυρία Γκροστέτ. Ναι, ξαναπαίρνω το λόγο γιατί ο συνάδελφος ο κύριος Πέτερλε ανησυχεί, διότι έχει την αίσθηση ότι οι ασθενείς παρόλα τις προσπάθειες που γίνονται από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τα μέσα που έχουν στη διάθεσή τους, ε, δεν είναι ακόμα σωστά πληροφορημένοι. Ρωτάει λοιπόν εάν μπορεί να υπάρξει μια πραγματική εκστρατεία ενημέρωση που θα απευθύνεται σε όλου του Ευρωπαίου πολίτε, όχι μόνο στου ε, ασθενεί, για να γνωρίζουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη οδηγία και ότι έχουν συγκεκριμένα δικαιώματα. Είναι αλήθεια ότι δεν γνωρίζουν τι περισσότερε φορέ τα δικαιώματά του, επομένω μπορούμε να κάνουμε πολύ περισσότερα και να του ενημερώσουμε ευρύτερα ή δυνατόν για να ενισχύσουμε την ενημέρωση των πολιτών καταρχάς, οι οποίοι δυστυχώς μπορεί μια μέρα να είναι ασθενείς που θα τους ενδιαφέρει το θέμα και να ε, μην βρεθούν και αυτοί λοιπόν σε αυτή τη ε, διαδικασία να ψάχνουν να βρουν τι θα γίνει. Θα είναι κρίμα δυο φορές. Ευχαριστώ πολύ. Άλλες ερωτήσεις προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Ο λόγος στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Πολύ καλή ερώτηση. Πώς μπορούμε να τα κάνουμε καλύτερα αυτά. Αναρωτιέμαι κι εγώ. Και στο Ευρωβαρόμετρο έχουμε την ερώτηση υπαριθμών 11. 11. Λοιπόν, ζητάμε από τους ερευνητές να συγκρίνουν τις γνώσεις που έχουν για το δικό τους το σύστημα και τις γνώσεις που διαθέτουν για τα δικαιώματα βάσει του ευρωπαϊκού συστήματος. Θα μπορούσα να χρησιμοποιήσω ίσως τη Γαλλία, παράδειγμα. Στη Γαλλία, για παράδειγμα, οι γνώσει των Γάλλων ασθενών και των οικογενειών τους είναι στο 68%. Δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά του βάσει του γαλλικού συστήματος υγεία. Ε, στα διασυνοριακά ε, δηλώνουν 15%. Ε, και μπορείτε να κάνετε μια σύγκριση να σας πω για τη χώρα μου, την Πολωνία. Στην Πολωνία οι ασθενείς και πάλι βάσει της μελέτης του Ευρωβαρομέτρου 44% δηλώνουν ότι γνωρίζουν το πολωνικό σύστημα υγεία και ένα ίδιο ποσοστό με τη Γαλλία, περίπου 14-15% δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα δικαιώματά τους για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας. Και αυτό που είναι ενδιαφέρον είναι ότι όταν ε, Είχαμε την εκστρατεία για την διασυνοριακή υγεία που έγινε σε τοπικό επίπεδο. Ε, διαπιστώνουμε ότι υπάρχει μεγάλη ροή ερωτήσεων από πολίτες, ε, πιθανούς ασθενείς, ακόμα και από ασθενείς και δεν μπορούσαν να απαντήσουν. Ε, ορισμένες φορές υπάρχουν εθνικά σημεία επαφής που δεν λαμβάνονται μια ερώτηση. Πώς μπορούμε λοιπόν να τα συμβιβάσουμε αυτά τα πράγματα μεταξύ των ε, πληροφοριών που παρέχουν τα κράτη-μέλη για αυτές τις δυνατότητες, που είναι φυσικά δικαίωμά τους και υποχρέωσή τους, ε, σε σχέση με την ανάγκη ε, να υπάρχει ενημέρωση σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Εμείς θεωρούμε ότι είναι πιο σημαντικό να βοηθούμε και να γίνουν αυτά σε ευρωπαϊκό επίπεδο, να υπάρχει μια μεγάλη ευρωπαϊκή εκστρατεία. πρέπει ίσως ε, ορισμένες φορές σε κάποιες χώρες να γίνει κατανοητό το δικό τους το σύστημα υγείας. Ε, για παράδειγμα υπάρχουν χώρες στις οποίες ε, δηλώνει ένα 24% ότι γνωρίζουν το σύστημά τους και ένα 12% εξ αυτών δηλώνουν ότι γνωρίζουν τα ευρωπαϊκά τους δικαιώματα. Είναι ένα δύσκολο ερώτημα. Κάποιοι λένε ότι δεν ξέρω καν το δικό μου το σύστημα, πώς να ξέρω το ευρωπαϊκό. Η κυρία Γκροστέτ. Νομίζω, δεν ξέρω, νομίζω ότι αυτή ήταν και ερώτηση του συναδέλφου Πέτερλε, ότι μια μεγάλη εξαρτή ενημέρωση των Ευρωπαίων πολιτών θα ήταν αυτό που είναι σημαντικό, διότι ε, φαίνεται ότι τα κράτη-μέλη δεν ενδιαφέρονται καθόλου και δεν θέλουν καν να ε, εφαρμοστεί η οδηγία για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας. Αυτό είναι το πρόβλημα. Πρέπει λοιπόν να ε, μπορέσουμε να ε, έρουμε τους δισταγμούς των κρατών μελών και αυτό φυσικά μπορεί να γίνει με κατάλληλη ενημέρωση και ενημέρωση όλων των Ευρωπαίων πολιτών και όχι μόνο των ασθενών. Των ε, Ευρωπαίων πολιτών που πρέπει να γνωρίζουν ότι υπάρχει μια οδηγία για τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας που μπορεί να τους δώσει ε, προγραμματισμένη θεραπεία σε άλλο κράτος μέλος ε, μπορούν να υποφαληθούν για διάφορους λόγους που γνωρίζουμε πολύ καλά και περιλαμβάνονται και στο κείμενο και γι' αυτόν ακριβώς το λόγο θα πρέπει να πάμε πέραν της διάθεση των κρατών μελών. Ευχαριστώ, Κύριε Σαλντεμός. Και εμένα με απασχολεί το ζήτημα λοιπόν της γνώσης που έχουν οι ασθενείς. Γιατί προφανώς εάν οι Ευρωπαίοι πολίτες δεν γνωρίζουν ακόμα τα, δικαιώματα τους ακόμα και στο ίδιο τους το κράτος μέλος, πώς ο, πιθανό είναι να γνωρίζουν τα δικαιώματα τους σε ευρωπαϊκό επίπεδο και να ρωτιέμαι, Για να πούμε κάποια στιγμή ότι καταφέραμε να υλοποιήσουμε πλήρως αυτό που θέλαμε, την οδηγία. Σε ποιο βαθμό θα πρέπει να υπάρχει αυτή η γνώση στους ασθενείς. Δηλαδή, αρκεί, μήπως αρκεί να γνωρίζουν απλώς οι ασθενείς ότι υπάρχει αυτή η δυνατότητα και μετά σε δεύτερο στάδιο, αν χρειαστούν ε, να εκμεταλλευτούν αυτήν την να αξιοποιήσουν αυτή τη δυνατότητα, τότε να τους παρέχετε επιπλέον πληροφόρηση για τις θεραπείες, τις διαδικασίες κτλ. αλλά με το ρυθμό που παρατηρείται αυτή τη στιγμή να υλοποιείται, να εφαρμόζεται η οδηγία. Πότε προβλέπετε, ποια χρονιά προβλέπετε ότι θα έχουμε φτάσει σε πλήρη εφαρμογή. Ευχαριστούμε, Επιτροπή. Πολύ καλή ερώτηση. Πραγματι, μετρώντας την ευαισθητοποίηση του κατά πόσον το κοινό γνωρίζει τη δυνατότητα αυτή ο Ευρωπαίος πολίτης είναι ένας τρόπος να γνωρίζουμε και κατά πόσον τελικά αυτή η οδηγία μπορεί να εφαρμοστεί. Εγώ είμαι αισιόδοξο και γενικά και εδώ. Πιστεύω ότι αν σιγά σιγά ξεκινήσουν οι πολίτες να χρησιμοποιούν αυτά τα δικαιώματά τους, θα γίνει περισσότερο γνωστό. Μπορούν επίσης να βοηθήσουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, αναδεικνύοντας τέτοιες ε, υποθέσεις. Στη Σλοβενία, για παράδειγμα, γνωρίζω ότι έγινε μια μεγάλη σημαντική δημόσια συζήτηση για το θέμα αυτό και διαπιστώνουμε ότι ένα αυξημένο ποσοστό Σλοβαίνων πολιτών γνωρίζει πια ποια είναι τα δικαιώματά του. Ότι γνωρίζει ότι έχει δικαιώματα σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Βεβαίω θα θέλαμε όλοι οι πολίτες να το γνωρίζουν. Αλλά σωστά επισημαίνεται ότι ε, οι πολίτες συχνά δεν γνωρίζουν καλά τα δικά του τα εθνικά συστήματα υγείας και ανάλογο είναι και το επίπεδο. Θα θέλαμε να είναι ανάλογο μάλλον το επίπεδο τη γνώση του για το ευρωπαϊκό σύστημα σε μικρότερες χώρες όπως η Μάλτα υπάρχει καλύτερη γνώση γιατί βεβαίως και για άλλους λόγους ε, αναγκάζονται να χρησιμοποιούν πιο συχνά τη διασυνοριακή παροχή υπηρεσιών υγείας. Για... Ε, βλέπουμε μια μικρή διαφορά στα ποσοστά μεταξύ εκείνων που γνωρίζουν που είναι επαρκώ ε, ενημερωμένοι για το εθνικό του σύστημα υγεία και για το 34% που γνωρίζει επαρκώ για το ευρωπαϊκό σύστημα υγεία. Επομένω πρέπει να σκεφτούμε ποιο είναι ο καλύτερο τρόπο για να προωθήσουμε αυτό το σύστημα. Βρισκόμαστε σε διάλογο και συζήτηση με τα κράτη-μέλη, αλλά είναι τα κράτη-μέλη που εφαρμόζουν την οδηγία. Και διαπιστώνουμε ότι κάθε κράτος μέλος την εφαρμόζει με διαφορετικό τρόπο. Ίσως αναγκαστούμε να προσφύγουμε στο δικαστήριο με διαδικασίες επί παραβάση. Το απέφχομαι, αλλά ίσως αυτό επίσης να αλλάξει τον τρόπο εφαρμογής της οδηγίας αλλά όλα τελικά εξαρτώνται από τα κράτη-μέλη και την διαθεσιμότητά τους να αξιοποιήσουν το σύστημα αυτό. Τουλάχιστον όμως με τα κράτη-μέλη με τα οποία συνεργάζομαι δεν διαπιστώνω να υπάρχει διάθεση να μπλοκάρουν το σύστημα. Ε, είναι διατεθειμένοι να δεχθούν ασθενή. Ευχαριστούμε. Μπορούμε να προχωρήσουμε στην επόμενη ερώτηση υπαριθμών 7. Δίνω και πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. έχουμε την διαδικασία παραβάσεων, η οποία είναι σημαντική. Είπα ήδη κατά την εισαγωγή μου ότι ξεκινήσαμε τη διαδικασία αυτή με 26 κράτη-μέλη. Της διαδικασίας παράβασης δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε με όλα αυτά τα κράτη-μέλη στο δικαστήριο. Έχουμε επικοδομητικό διάλογο και προσπαθούμε να κατανοήσουμε τις νομικές διατάξεις, καθώς και πώς εφαρμόζονται στην πράξη τα συστήματα αυτά. Το θέμα λοιπόν είναι πώς, έχουν μεταφερθεί, πώς έχει μεταφερθεί η οδηγία στη νομοθεσία των κρατών μελών. Να σας δώσω κάποια παραδείγματα, διότι δεν θέλω να αναφερθώ σε όλα τα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη έχουν ιδιαίτερα πολύπλοκο σύστημα προηγούμενης έγκρισης. Θέλουμε να το καταλάβουμε καλύτερα, διότι έχουν δικαίωμα να εφαρμόζουν ένα τέτοιο ε, σύστημα, αλλά μήπως είναι τρόπος ε, να ε, κλείσουν την πρόσβαση στη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Άλλα κράτη έχουν χαμηλότερο ποσοστό επιστροφής. Βρισκόμαστε σε διάλογο με αρκετά κράτη-μέλη. Καταλαβαίνουμε ότι τα ποσοστά αυτά συνδέονται με ένα σωρό συστήματα του παρελθόντος. Και τέλος, θέλουμε να καταλάβουμε, διότι εάν είναι ιδιαίτερα επαχθές το σύστημα, οι ασθενείς δεν έχουν την απαραίτητη γνώση, δεν έχουν πάντα δικηγόρους μαζί τους για να εποφεληθούν από τη διασυνοριακή υγειονομική περίθαλψη. Τέλος, θέλουμε να δούμε πώς λειτουργεί στην πράξη το σύστημα, τι κάνει ο ασθενή δηλαδή για να υποφεληθεί από το σύστημα αυτό. Αυτό είναι το σχέδιο μα. Ευχαριστώ. Η κυρία Γκροστέτ. Ναι, οι εξηγήσει που μας δόθηκαν είναι πάρα πολύ ενδιαφέρουσέ βεβαίω. Κατανοούμε πάρα πολύ καλά ε, τα θέματα αυτά. Πάντα μιλάω εξ ονόματο του κυρίου Πέτερλε, αλλά υπάρχει μια πραγματική ανησυχία. Να δούμε αν μπορούμε να ελέγξουμε τη μεταφορά της οδηγίας ε, στα 28 κράτη-μέλη, αλλά κατόπιν θα υπάρχει και το θέμα της σωστής εφαρμογής ε, αυτής της οδηγίας. Ε, Αυτή τη στιγμή τη μεταφέρουμε. Νομίζω ότι ο συνάδελφος ήθελε να ξέρει εάν στην περίπτωση που τα δικαιώματα των ασθενών ε, σαφώς παραβιάζονται ή στην περίπτωση στην οποία διαπιστώσουμε ότι υπάρχουν πραγματικά περιτά εμπόδια τα οποία ε, θέτουν τα κράτη-μέλη, θα υπάρχει διαδικασία επιπαραβάση ε, ή κάποιες κυρώσεις ε, κατά των κρατών μελών ε, οι οποίοι δεν θα τηρούν τα όσα προβλέπονται. Νομίζω ότι αυτό έχει σημασία όχι μόνο για την ποιότητα του κειμένου αλλά και τη σωστή εφαρμογή. Ξέρουμε τι προβλήματα υπήρχαν για την έγκριση της οδηγίας. Θα πρέπει λοιπόν να επαγρυπνούμε στη συνέχεια. Πώς θα φροντίσετε να τα παρακολουθήσετε όλα αυτά και σε περίπτωση που ε, παραβιάζονται τα δικαιώματα των ασθενών πώς θα τιμωρείτε. Ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Όχι. Ωραία λοιπόν ο λόγος των Κομισιόν. Λοιπόν, όπως σας είπα, έχει γίνει ο έλεγχος της πληρότητας. Όλα τα κράτη-μέλη έχουν εφαρμόσει, κάποια θα αργήσουν λίγο σε κάτι, αλλά ε, έχει γίνει αυτός ο έλεγχος του κατά πόσο είναι πλήρη τα πράγματα και ε, βεβαίως στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπάρχει ένα πλήρες οπλοστάσιο το οποίο θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε αν χρειαστεί. Αυτή τη στιγμή όμως, επειδή η οδηγία αυτή, όπως γνωρίζουμε, είναι πολύ περίπλοκη, διότι έχουμε να κάνουμε με 28 διαφορετικά συστήματα. Επομένως πρέπει να ε, παραπέμπουμε θέματα στα κράτη-μέλη, θέλουμε να κατανοήσουμε πώς ε, γίνονται κάποια πράγματα και επίσης μην ξεχνάμε ότι ε, οι ασθενείς έχουν κάθε δικαίωμα προσφυγή στο δικαστήριο. Ε, κατά τη διαπραγμάτευση συζητήσαμε ότι η χειρότερη περίπτωση θα είναι να έχουμε πάρα πολλές υποθέσεις στο δικαστήριο. Ε, και αυτή η οδηγία ξεκίνησε από τις πολλές προσφυγές. Σαφώς και υπάρχουν δικαιώματα για τις ασθενείς ε, και εγώ ξέρω μια χώρα στην οποία προσέφυγαν οι ασθενείς πριν από την μεταφορά της οδηγίας και ρώτησαν γιατί δεν ε, μεταφέρει την οδηγία η χώρα μου και το Εθνικό Δικαστήριο τους έδωσε δίκιο. Επομένως, ελπίζουμε ότι αυτή τη στιγμή θα μπορέσουμε να δούμε πόσο χρόνο χρειαζόμαστε και πόσο θα χρειαστεί, ώστε πραγματικά να κατανοήσουμε αυτή τη στιγμή, προσπαθούμε να καταλάβουμε, διαπραγματευόμαστε, προσπαθούμε να εξηγήσουμε ένα τον άλλον, αλλά σίγουρα θα περάσουμε και στο επόμενο στάδιο κάποια στιγμή. Ευχαριστώ πολύ. Να πάμε στην επόμενη ερώτηση, στην ημερήσια διάταξη. Πρόκειται για την υπαριθμό 8, προστασία δεδομένων και ασφάλεια δεδομένων και προστασία. Ο λόγος στην Κομισιόν. Συζητάμε λοιπόν για την ανταλλαγή ε, ευαίσθητων προσωπικών δεδομένων, ε, δεδομένων που αφορούν σε ασθενείς. Βεβαίως και γίνεται πλήρως σεβαστή η οδηγία για την προστασία των προσωπικών δεδομένων και ιδιαίτερα στον τομέα της υγείας. Προσπαθούμε να χρησιμοποιήσουμε το πληροφοριακό σύστημα ε, για την ενιαία αγορά, το IMIS που δίνει τη ε, δυνατότητα ανταλλαγής με, με ασφάλεια πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών. Αυτές είναι οι συνθήκες επί τους οποίες εργοζόμαστε. Σιγά σιγά δημιουργείται και μια νέα πλατφόρμα, ε, ένα νέο πληροφοριακό σύστημα χρησιμοποιώντας χρηματοδότηση από το χρηματοδοτικό εργαλείο συνδέοντας στην Ευρώπη, το Connecting Europe, που θα δώσει τη δυνατότητα διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων των συστημάτων υγείας στα διάφορα κράτη-μέλη. Ε, προβλέπουμε το νέο σύστημα αυτό να ε, ξεκινήσει να λειτουργεί από το 2018. Τότε να δίνουμε τη δυνατότητα στα κράτη-μέλη που το επιθυμούν να το αξιοποιήσουν. Ο Πρόεδρος, σας ευχαριστούμε. Για Κάντεμπακ, αν δεν κάνω λάθο. όχι, δεν θέλετε το λόγο. Μήπω κάποιο άλλο συνάδελφο θέλει να λάβει το λόγο επί αυτού του ερωτήματο. Όχι, άρα μπορούμε να περάσουμε στο επόμενο. Ένατο ερώτημα. Μελλοντικά ε, μέτρα, μέτρα που θα ληφθούν στο μέλλον. Μιλάμε για τη διασυνοριακή συνεργασία και θα πρέπει πρώτα να σκεφτούμε πώς αντιλαμβανόμαστε την διασυνοριακή συνεργασία. Μπορεί να πραγματοποιείται μεταξύ δύο περιφερειών. Για παράδειγμα, έχουμε τη συνεργασία μεταξύ ε, Ισπανίας και Γαλλίας στα Πυρηναία, έχουμε μεταξύ Βελγίου και Λουξεμβούργου, ανάμεσα στις κάτω χώρες ε, και τη Γερμανία. Συμφωνία στο Καλέ. Έχουμε λοιπόν διάφορες ε, γειτονικές περιφέρειες. Μετά έχουμε διαπεριφερειακή συνεργασία, όπου βλέπουμε δύο περιφέρειες μη γειτονικές, να συνεργάζονται. Είδαμε για παράδειγμα τέτοιο πρόγραμμα συνεργασίας ανάμεσα στη Σκωτία και την Νότια Ισπανία που απέχουν αρκετά. Και έχουμε και την διεθνική συνεργασία, για παράδειγμα την Μεσογειακή, όπου συμμετέχουν η Ελλάδα, η Κροατία, η Ιταλία, η Ισπανία ή την περιφέρεια του Δούναβη. Έχουμε λοιπόν διάφορες τέτοιες περιοχές όπου συχνά η υγεία αποτελεί μέρος της συνολικής συνεργασίας στηρίζουμε τις προσπάθειες αυτές, προσπαθούμε να υποστηρίξουμε τη συνεργασία με τις βέλτιστες πρακτικές, χαρτογραφούμε τη συνεργασία με τα διαρθρωτικά ταμεία ή μέσω του Ίντερεγ. Και πιστεύουμε ότι η συνεργασία αυτή είναι δυνατή μόνο όταν υπάρχει βούληση από πλευράς ε, της τοπικής ε, ε, διοίκησης ε, με την ευλογία της κυβέρνησης. Χρειάζονται και οι δύο αυτοί παράγοντες. Επίσης, ζητάμε από το πάνελ εμπειρογνωμόνων μας ε, να γνωμοδοτήσει σχετικά με τις συνεργασίες αυτές. Ζητήσαμε να εντοπίσουν πέρσι ποια είναι τα συγκεκριμένα εμπόδια σε τέτοιου τύπου συνεργασία. Πώς μπορούν να εξοικονομηθούν πόροι, ε, πώς μπορεί να αποφευθεί η δημιουργία νέων υποδομών εάν δεν ε, είναι απαραίτητες, ε, πώς μπορούμε να σκεφτούμε με τρόπο καινοτόμο. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Κάτενμπαχ θέλει να απαντήσει, όχι. Ωραία, σας ευχαριστώ πολύ. Ήταν πολύ σαφής η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο θέμα αυτό. Πάμε στην ερώτηση 10, αξιολόγηση των υπαρχόντων συστημάτων. Το δίνω, δίνω πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Είδατε τις ε, Είδατε την επιστολή του ε, Επιτρόπου μου. Του ζητήθηκε να αναπτύξει ένα σύστημα το οποίο προσπαθήσαμε να υπονοήσουμε σε συνεργασία με τους εμπειρογνώμονες των κρατών μελών. Ο πρώτος τομέας με τον οποίο ασχοληθήκαμε ήταν η ποιότητα της υγειονομικής περίθαλψης και μόλις ολοκληρώσαμε την έκθεση η οποία παρουσιάστηκε στα κράτη-μέλη αρχές Φεβρουαρίου εδώ στις Βρυξέλλες. Ελπίζουμε να δημοσιευτεί εντός του επόμενου μήνα. Πιστεύουμε ότι ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η δουλειά αυτή. Έδειξε πόσο δύσκολο είναι να μετρηθούν και να συγκριθούν πράγματα μη μετρήσιμα και μη συγκρίσιμα. Προσπαθήσαμε να συνεργαστούμε στενά με τον ΩΣΑ και το παρατηρητήριο για τις ε, υγειονομικές πολιτικές εδώ στις Βρυξέλλες. Επίσης, καλέσαμε τους εμπειρογνώμονές μας, στους οποίους ήδη αναφέρθηκα, να του ζητήσαμε να εξετάσουμε το θέμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας, διότι αυτό είναι πάντα το δύσκολο θέμα για ό,τι έχει να κάνει με την ιστορία των κρατών μελών. Πιστεύουμε ότι έγινε πολύ θετικά αποδεχτή. Είχαμε πολλές παρατηρήσεις και στη δημόσια διαβούλευση και εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε το θέμα αυτό σε μια συνεδρίαση. Και Είχαμε και την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που δημοσιεύθηκε το 2014, όπου αναφερόμαστε στα συστήματα υγειονομικής περίθαλψης. Προσπαθήσαμε λοιπόν ε, να παράσχουμε βοήθεια και να μπορέσουμε να απαντήσουμε στις ερωτήσεις. Ευχαριστούμε. Υπάρχει κάποιος συνάδελφος που θέλει να θέσει κάποιο ερώτημα. Όχι. Αν όχι, ας περάσουμε στο επόμενο. Ε, κέντρα αριστείας. Πρόσωπος της Επιτροπής. Και πάλι έχει με άλλο ενδιαφέρον το ερώτημα αυτό. Ήδη ε, ανέφερα το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Αναφοράς ως ένα σύστημα ενίσχυσης της ευρωπαϊκής συνεργασίας. Τα κέντρα αριστείας είναι μια ε, λογική, μια έννοια η οποία χρησιμοποιείται στις επιστήμες, στην ακαδημαϊκή έρευνα και στην κλινική πρακτική. Αυτό το γνωρίζουμε από διάφορα κράτη-μέλη. Εμείς επιδιώκουμε να προσκαλέσουμε ε, και να ζητήσουμε από όλα τα κέντρα αριστείας, δηλαδή από όλα τα κέντρα ε, που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της ε, έρευνας και της περίθαλψης στον τομέα της υγείας, να συνεργαστούν. Το ζήτημα δεν είναι τόσο πολύ η αριστεία όσο η διάθεση συνεργασίας. Και ελπίζω ότι θα την ενισχύσουμε αυτή τη διάθεση συνεργασία, γιατί έτσι θα υποφεληθούν οι ασθενεί όχι μόνο από ένα κέντρο εξαιρετικό στην Ιταλία, για παράδειγμα, αλλά επίση από τη συνεργασία αυτού του κέντρου με ένα άλλο κέντρο, για παράδειγμα, στη Γαλλία ή αλλού. Δηλαδή, οι ασθενεί θα υποφεληθούν από το γεγονό ότι συγκεντρώνεται και μοιράζεται η γνώση αναμεταξύ όλων των μελών του δικτύου. Και αυτή η ανταλλαγή των επιστημονική γνώση είναι ο τομέα στον οποίο η Ευρωπαϊκή Ένωση φέρνει την προστιθέμενη αξία τη. έχουμε στο, στην Ιταλία, επειδή η Ιταλία ε, είναι πολύ μπροστά σε αυτόν τον τομέα. Έχει δημιουργήσει ένα ε, σύστημα. Ε, στην Ιταλία, όπως γνωρίζετε, οι ε, νομοί έχουν μεγάλη σημασία και ε, υπάρχει μια σχετική αυτονομία. Επομένως, ευελπιστούμε ότι πολλά και διαφορετικά κέντρα της Ιταλίας θα συμμετάσχουν τελικά στο ευρωπαϊκό σύστημα. Πάντως προσπαθούμε αυτή η πρωτοβουλία να ξεκινήσει από τα κάτω, από, τις, τα κατατόπους ερευνητικά κέντρα. Ευχαριστούμε κύριο Πετιτσίνη ή από κάποιον άλλο συνάδελφο προς την Επιτροπή. Δεν έχουμε κάποιο ερώτημα. Μπορούμε να περάσουμε στο, στα επόμενες δύο μάλλον ερωτήσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να τις δούμε μαζί. Ο εκπρόσωπος της Επιτροπής. Λοιπόν, η πρώτη ερώτηση αφορά την εφαρμογή και τα προσκόμματα για την ε, ελεύθερη κυκλοφορία των ασθενών και νομίζω ότι το έχουμε συζητήσει αυτό και ήταν σαφές ότι Αυξάνεται η ενημέρωση, όπως γίνεται στον καταναλωτικό κόσμο, τα δικαιώματα των ασθενών πρέπει να γνωστοποιηθούν και μετά να μπορεί κάποιος να τα ασκήσει φυσικά. Και αυτή είναι η πρώτη σημαντική ε, στιγμή για τα όσα κάνουμε και από εκεί και πέρα θα πρέπει να δούμε στη ε, διαδικασία συμμόρφωσης με τα κράτη-μέλη, θα δούμε τι προσκόμματα υπάρχουν ε, για την όλη ελεύθερη κυκλοφορία. Και νομίζω ότι η απάντηση είναι η ίδια ε, με την ερώτηση που συζητήσαμε και προηγουμένως. Όσον αφορά τη δεύτερη, για αυτή τη δομή του θεματοφύλακα, στις συζητήσεις μας και στο κείμενο της οδηγίας συμφωνήσαμε ότι ο τρόπος ε, με τον οποίο θα υπάρχει αυτή η προστασία του gatekeeper στα κράτη-μέλη θα πρέπει να παραμείνει. Εάν χρειάζεται αναφορά, ε, παραπομπή μάλλον ε, για ακριβή θεραπεία στη χώρα καταγωγής, θα πρέπει να συνεχίσει με αυτόν τον τρόπο. Τα κριτήρια δεν θα πρέπει να διαφέρουν φυσικά και παρεπιπτόντος είναι και ένας από τους τομείς που θα θέλαμε να εξετάσουμε περαιτέρα. Εάν ε, στη μεταφορά τους τα κράτη-μέλη μήπως ε, διεύρυναν τα κριτήρια και πρόσθεσαν πολλά περισσότερα για αυτούς που θέλουν να πάνε στο εξωτερικό. Ε, Δηλαδή μια χώρα που καθορίζει τα κριτήρια για την εξειδικευμένη θεραπεία δεν θα πρέπει να προσθέτει επιπλέον ε, κριτήρια για την ε, μεταφορά του ασθενού στο εξωτερικό από όσα ε, προβλέπονται σε εθνικό επίπεδο. Όπως σας είπα ήδη, εάν θεωρήσουμε ότι δεν λειτουργεί αυτό όπως θα έπρεπε να λειτουργεί, θα υπάρξουν διαδικασίες επί και θα τα συζητήσουμε αυτά παρετέρω. Ευχαριστώ πολύ. Ο λόγος στην κυρία Σαλτεμός. Ευχαριστώ πολύ. Είναι αλήθεια ότι ήδη έχουμε συζητήσει το θέμα της ευαισθητοποίησης των ασθενών. Έχω όμως μια πιο γενική ερώτηση, διότι ένα θέμα είναι η ευαισθητοποίησή τους, άλλο θέμα είναι ότι είναι πολύ δύσκολο να εφαρμοστεί πλήρως η οδηγία αυτή και ότι υπάρχουν κάποια εμπόδια. Έχω λοιπόν ερώτηση. βλέπετε να υπάρχουν μοτίβα όσον αφορά τα εμπόδια. Υπάρχουν, ε, για παράδειγμα, κράτη-μέλη με ε, υψηλότερη φορολόγηση που να ε, εμποδίζουν τη διασυνοριακή περίθαλψη ή υπάρχει διαφορά βορρά και νότου ή έχουμε 28 διαφορετικά συστήματα. Και μία ερώτηση ακόμα. Πότε πιστεύετε ότι θα έχουμε ένα πλήρως λειτουργικό σύστημα για τη διασνοριακή υγειονομική περίθαλψη σε 5 χρόνια, σε 10 χρόνια. Πότε πιστεύετε ότι θα λειτουργεί πραγματικά καλά το σύστημα. Σας ευχαριστώ πολύ. Δεν ξέρω αν υπάρχουν άλλες ερωτήσεις. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Θα αναφερθώ και πάλι πρώτα στην μελέτη του Ευρωβαρόμετρου. Περίπου το 30% των ερωτηθέντων είπαν ότι θα θέλαμε να εξετάσουμε τη δυνατότητα. Νομίζω ότι αυτό είναι αρκετά υψηλό ποσοστό. Δεν γνωρίζουμε αν θα θέλανε να πάνε επειδή δεν μπορούν να λάβουν περίθαλψη στην πατρίδα τους ή αν το θεωρούν ευκαιρία. Διότι γενικά ξέρουμε ότι όλοι προτιμούν να λαμβάνουν υγειονομική περίθαλψη όσο γίνεται πιο κοντά στο σπίτι τους. Το ότι είμαι διατεθειμένος να πάω δεν σημαίνει απαραίτητα ότι θα επιλέξουν ε, τη δυνατότητα αυτή όταν βρεθούν στην κατάσταση να τη χρειάζονται. Εάν πάω λοιπόν στο εξωτερικό, τι είδους καθεστώς θα αντιμετωπίσω, μπορώ να λάβω υπηρεσίες στη δική μου γλώσσα. αν μιλάει κανείς μια μεγάλη γλώσσα, πιθανότατα να έχει καλύτερη πρόσβαση. Αλλά υπάρχουν και κέντρα που ειδικεύονται στην πολυγλωσία. Ιδιαίτερα όσον αφορά χειρουργικές επεμβάσεις που μπορούν να προγραμματιστούν ε, εκ των προτέρων ε, υπάρχει αυτή η δυνατότητα. Επίσης, ε, κάποιοι ασθενείς άρχισαν να ζητούν ε, μετάφραση ε, του φακέλου τους, ο οποίος μπορεί να είναι μία ή δύο σελίδες, μπορεί όμως να είναι και 30 ή 40, 100 σελίδες. Σκεφτείτε λοιπόν το κόστος τέτοιας εξειδικευμένης μετάφρασης. Θα θέλαμε λοιπόν να εξετάσουμε αυτές τις πρακτικές. Απ' την άλλη βλέπουμε και νέα φαινόμενα. βλέπουμε να, εμφανίζονται διαμεσολαβητές που θέλουν να βοηθήσουν. Δεν έχουμε πάντα τις απαραίτητες γνώσεις, ζητάμε από τα κράτη-μέλη να μας εξηγήσουν πώς έχει η κατάσταση. Άλλο παράδειγμα δυσκολιών. Συνδέεται με την κοινή γνώμη. Υπάρχει ο λεγόμενος τουρισμός ε, στον τομέα της υγείας. Συχνά λοιπόν ακούμε να συζητιέται ο τουρισμός της υγείας και όλες οι σχετικές υπηρεσίες όπου μπορεί το ποσοστό επιστροφής ε, να είναι σχεδόν μηδενικό όπως ε, είναι η πλαστική χειρουργική ή οι οδοντιατρικές εργασίες. Συχνά όμως ε, η πλαστική ε, χειρουργική ε, είναι απαραίτητη σε ανθρώπους με κάποιο πρόβλημα υγείας. Και τέλος, με ρωτάτε πόσος χρόνος απαιτείται. Νομίζω ότι εξαρτάται από όλους μας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καταβάλει κάθε προσπάθεια και τα κράτη-μέλη για την εφαρμογή της οδηγίας αυτής εντός του πλαισίου τους και οι επαγγελματίες στον χώρο της υγείας και οι ασθενείς ε, νομίζω επίσης ε, πως κινούνται προς αυτή την κατεύθυνση. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μπορούμε να κλείσουμε το θέμα αυτό της εφαρμογή τη νομοθεσία σχετικά με την υγεία. Ευχαριστώ θερμά την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Μπορούμε τώρα να περάσουμε στο επόμενο θέμα τη ημερήσιας διάταξη. Η επιδημία του ιού Ζήκα. Το χειροκρότημα ήταν για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, νομίζω. Έχουμε λοιπόν πρόταση ψηφίσματος και θα ακούσουμε τους συνεισηγητές, την κυρία Σράγερ Πίρικ. Σε ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Προφανώς ε, πρέπει να ξεκινήσουμε την καταπολέμηση του ιού Ζήκα πριν να ξεφύγει η κατάσταση από κάθε έλεγχο. Δεν είναι μόνο το ζήτημα ε, των κουνουπιών, πώς θα, θα περιορίσουμε. Χρειάζεται λήψη επιγόντων, επιγόντως μέτρων. Η Κομισιόν εκτιμά το κόστος της καταπολέμησης της επιδημίας στα 10 εκατομμύρια. Ε, εγώ πιστεύω ότι μπορεί να είναι πολύ υψηλότερο, ε, ιδίως ε, εάν χρειαστεί έρευνα για ένα εμβόλιο να χρηματοδοτηθεί έρευνα για ένα εμβόλιο στο πλαίσιο πιθανώ τη στρατηγική Ευρώπη 2020. Πρέπει να κινητοποιηθούμε πριν να φτάσει η επιδημία να επηρεάζει του Ευρωπαίου στην Ευρώπη. Γνωρίζουμε ότι χρειάζεται ε, επιτήρηση, παρακολούθηση της εξέλιξης, της διά, ε, εξάπλωσης του ιού και να δοθούν τα απαιτούμενα ε, εργαλεία και οι στην Επιτροπή για να παρακολουθεί ε, τις μεταφορές φορτίων, ε, ταξιδιωτών επίσης με αεροπλάνα από τις πληγήσεις περιοχές. Γνωρίζουμε ότι ένα από τα συμπτώματα, ένα, μάλλον ένα, ένα από τα αποτελέσματα του ιού είναι η μικροκεφαλία όταν και αυτές οι γενετικές ανομαλίες. Είναι πραγματική τραγωδία από ανθρώπινη πλευρά, την οποία πρέπει να προσπαθήσουμε στο μέτρο του φυκτού να αποφύγουμε και να περιορίσουμε. Η πρωτοβουλία λοιπόν ψηφίσματος που προτείνουμε έχει την υποστήριξη όλων των πολιτικών ομάδων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Νομίζουμε, νο, θεωρούμε ότι σε αυτό το θέμα μπορούμε όλοι ενωμένοι να ε, εκφραστούμε ανεξαρτήτως διαφορών πολιτικών, γιατί ε, πρόκειται για την υγεία και τη ζωή ε, εκατομμυρίων γυναικών εγγύων σε ολόκληρη την Ευρώπη. Ευχαριστώ, ο κύριος Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζω ότι τα στοιχεία που έχουμε αποτελούν πολύ καλή βάση για τη συζήτηση πάνω στο θέμα αυτό. Έχουμε παραπέμψει το θέμα στην ε, Ειδική Επιτροπή. Θέλουμε λοιπόν να εξετάσουμε προσεκτικά το θέμα και όχι απλά να έχουμε ε, μία υψηλών τόνων συζήτηση στην Ολομέλεια. Μας ενδιαφέρει λοιπόν η έρευνα και η ανάπτυξη. Υπάρχουν ε, δυνατότητες εντός ε, του εβδόμου προγράμματος, ε, προγράμματος πλαισίου και του προγράμματος Ευρώπη 2020 να ασχοληθούμε με το θέμα και όπως ήδη υπόθηκε θα πρέπει να περιορίσουμε την εξάπλωση του ιού και γι' αυτό θα πρέπει να γνωρίζουμε πώς μεταδίδεται. Πολύ συγκεκριμένα, διότι δεν έχουν ερευνηθεί ακόμα και οι τελευταίες λεπτομέρειες. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να πραγματοποιηθεί η συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών, διότι λόγω της ε, παγκοσμιοποίησης Ενδιαφέρον είναι λοιπόν να δούμε πώς έχει εξαπλωθεί ο ιός και πώς μπορούμε να περιορίσουμε την περαιτέρω εξάπλωσή του. Νομίζω ότι έχουμε ένα καλό ψήφισμα το οποίο μπορούμε να υιοθετήσουμε και το οποίο περιέχει και κατευθυντής γραμμές για το πώς μπορούμε να κινηθούμε. Έχει οδηγήσει ο ιός αυτός σε μικροκεφαλία και δυσμορφία σε βρέφη. Θα πρέπει λοιπόν να εξετάσουμε πού οφείλονται ε, αυτές οι περιπτώσεις. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φαρία, εκ μέρους των Φιλελευθέρων. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η συγκεκριμένη ανησυχία ε, που ε, μας οδηγεί στην ε, ταχεία έγκριση για τα μέτρο για την ε, με βρίσκει σύμφωνο με τα όσα είπε ο κύριος ε, Γκρότε. Είναι πάρα πολύ σοβαρή η κατάσταση και τώρα που πλησιάζει η Άνοιξη και το καλοκαίρι, αν δεν είμαστε κατάλληλα προετοιμασμένοι, είναι πάρα πολύ πιθανό και πολύ εύκολο να φτάσει ο ιός στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τα νέα είναι όλο ένα και πιο ανησυχητικά. υπήρξε αυτή η ραγδαία αύξηση των περιστατικών όχι μόνο στην Βραζιλία αλλά και στη Βενεζουέλα και στην Κολομβία. Γνωρίζουμε ότι όπως επισημάθηκε εδώ σε αρκετές περιπτώσεις ότι ο ιός μεταδίδεται όχι μόνο από ε, τσίπη αλλά και από μέσω της σεξουαλικής επαφής ε, και μέσω μετάγγισης αίματος. Ε, σήμερα ήταν εδώ η κυρία Αμών από το Κέντρο Πρόληψης νόσους, Νόσων και την προηγούμενη εβδομάδα ο κύριος Μπερτόλη από την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Και αυτό νομίζω ότι αντανακλά και τη σημασία που έχει το θέμα αυτό για όλους. Πρέπει να δράσουμε τώρα και εγώ θα ήθελα να συγχαρώ τους ε, εισηγητές του ψηφίσματος. Ε, έχουμε καταφέρει να καταλήξουμε σε συνένεση μεταξύ μας ε, για το κείμενο και θέλουμε πραγματικά να τεθούν σε επιφυλακή τα ευρωπαϊκά όργανα για την απειλή αυτή και να μπορέσουμε να καταπολεμήσουμε την πιθανότητα επιδημίας και να ευαισθητοποιήσουμε τους Ευρωπαίους πολίτες. όπως πολύ σωστά ακούστηκε και σήμερα νωρίτερα, θα πρέπει να ε, υπάρξουν και κάποια διδάγματα από την επιδημία του έμπολα που έφτασε σε μια στιγμή ε, το 2014. Πρέπει λοιπόν να δράσουμε πολύ πιο γρήγορα και πιο αποτελεσματικά από ό,τι τότε, διότι αυτό είναι ένα ε, σημαντικό θέμα για την υγεία όλων. Θεωρώ ότι είμαστε στη σωστή κατεύθυνση και ελπίζουμε ότι από εδώ και πέρα και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορέσει να πει κάτι επί του ζητήματος και θα μελετήσει εις βάθος ε, το ζήτημα αυτό και να φτάσουμε και στην πλήρη εξάλληψη του ιού. Ευχαριστώ κύριε Σπιέκα. Θα πρέπει να στηρίξουμε το ψήφισμα αυτό και ήρθε η ώρα να αναλάβουμε δράση. Ε, είδαμε άλλωστε παρόμοιες καταστάσεις στην περίπτωση του ιού έμπολα. Θα πρέπει να λάβουμε υπόψη μας και τις αναλογίες, ε, διότι ο ιός έπολα αποτελούσε πολύ μεγαλύτερη απειλή. Σημαντικό όμως είναι να δραστηριοποιηθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Δεν χρειάζεται κάθε φορά να επινοούμε νέες διαδικασίες. Υπάρχουν πολύ κίνδυνοι στη φύση για τους ανθρώπους ε, και ίσως θα ήταν χρήσιμο να αναπτύξουμε σχετικές διαδικασίες. Να εξετάσουμε, για παράδειγμα, την ε, δυναμική της εξάπλωσης μιας επιδημίας. Αυτό είναι σημαντικό για την προστασία της υγείας των Ευρωπαίων πολιτών. Σημαντικό είναι να παρασχεθεί και η οικονομική υποστήριξη, ιδιαίτερα στους τόπους εμφάνισης του ιού. Στις μέρες μας ε, μιλάμε για τις επιπτώσεις του ιού Ζήκα στους Ευρωπαίους πολίτες. Δεν υπάρχει άμεση απειλή, υπάρχουν κάποιες ανησυχίες και ενημερώνεται ο κόσμος ε, σχετικά με το πώς θα πρέπει να κινηθεί. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε τι μέτρα πρόληψης θα πρέπει να εφαρμόσουμε. Ε, στηρίζω το σχέδιο ψηφίσματος. Ευχαριστούμε κυρία Κανιάτσινα. Συμφωνώ και εγώ λοιπόν με τους ε, συναδέλφους που συνέταξαν αυτό το ψήφισμα. Είχαμε πολύ καλή συνεργασία και πιστεύω ότι καταλήξαμε σε ένα ε, κείμενο το οποίο καλύπτει όλα τα σημαντικά ζητήματα που άπτονται του ιού ζήκα ε, της επιδημίας αυτής. Διαπιστώνουμε ότι νέα στοιχεία ε, έρχονται στη δημοσιότητα, τα μαθαίνουμε σιγά σιγά για τον τρόπο εξάπλωσης του, ιού, ε, για την μικροκεφαλία. Ε, ίσως να έχουν, να, έχουν υπάρξει μεταλλάξεις, να έχουν υπάρξει ε, αλλαγές στον τρόπο με τον οποίο λειτουργεί αυτός ο ιός τα τελευταία δέκα χρόνια. έχει τεθεί επίσης το ερώτημα εάν η μικροκεφαλία προκλήθηκε από τον Ιωζίκα ή από τη χρήση εντομοκτώνων. Και αυτό πρέπει να μας απασχολήσει, πρέπει να υπάρξει μια απάντηση γιατί ανησυχούν και οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και στην πρωινή μας συζήτηση αναφέρθηκε ότι έχουμε στη διάθεσή μας το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νόσων, το οποίο πριν ξεκινήσει αυτή η επιδημία που ε, έχουμε σήμερα, η επιδημία του, του ε, ΣΥΚΑ, είχε ξεκινήσει να δραστηριοποιείται, είχε ε, διοργανώσει εκστρατείες ευαισθητοποίησης, προσπαθώντας να ενημερώσει τους Ευρωπαίους πολίτες για τους κινδύνους. Νομίζω ότι αυτό καταδεικνύει τη σημασία που έχουν τέτοιου τύπου ε, υπηρεσίες σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μας δίνουν τη δυνατότητα να ανταποκρινόμαστε σε κρίσεις ε, σε επίπεδο της Ευρωπαϊκής Ένωσης πολύ πιο γρήγορα. Υποστηρίζουμε λοιπόν και εμείς το ψήφισμα, το οποίο θεωρούμε ότι είναι το πρώτο βήμα βέβαια, θα χρειαστούν και άλλα μέτρα και από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης Νόσων. Γνωρίζουμε ότι ο ιός αυτός ε, έχει εξαπλωθεί σε περιοχές προς τις οποίες πρόκειται να ταξιδέψει μεγάλος αριθμός Ευρωπαίων πολιτών σύντομα, όταν έρθει το καλοκαίρι. Ε, και θα πρέπει να είναι ε, ενήμεροι οι πολίτες για το πώς μπορούν να ε, προστατευτούν, να προετοιμαστούν, έτσι ώστε να αποφύγουμε περαιτέρω εξάπλωση του ιού. Σας ευχαριστώ, ευχαριστώ και τους συναδέλφους για την καλή συνεργασία που είχαμε στην κατάρτιση του ψηφίσματος. Ο Πρόεδρος, ευχαριστούμε. Η κυρία Χάουσλιν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να τονίσω αυτό που είπαν ο και οι προλαλήσαντες. Είναι σημαντικό να έχουμε κοινή βάση κατά τις ε, μελλοντικές μας δράσεις. Θα πρέπει να εξετάσουμε πολύ προσεκτικά τις ε, αιτίες εμφάνισης του ιού. Δεν εμφανίστηκε από τη μία μέρα στην άλλη. Χρειαζόμαστε περισσότερες γνώσεις λοιπόν. Η γρήγορη εξάπλωση δείχνει επίσης ότι δεν ε, θα περιοριστεί ε, στο νότιο ημισφαίριο η εξάπλωση κάποια στιγμή θα εμφανιστεί και στην Ευρώπη. Θα πρέπει λοιπόν ε, να το θεωρήσουμε παγκόσμιο πρόβλημα και όχι μόνο του νότου. Υπάρχουν ε, πολλά ερωτήματα που δεν έχουν ξεκαθαριστεί. Υπάρχει άλλωστε και η υποψία ότι η εξάπλωση του ιού, μάλλον ε, της μικροκεφαλίας, ε, συνδέεται με συγκεκριμένο εντομοκτόνο. Το θέμα είναι πώς μπορούμε να βοηθήσουμε τους ανθρώπους επιτόπου, πώς μπορούμε να λάβουμε μέτρα που να βοηθήσουν τους ανθρώπους, για παράδειγμα, να μοιράσουμε κουνουπιέρες. Θα πρέπει επίσης να καταστήσουμε σαφές ότι δεν μπορούμε ε, ε, να εξαφανίσουμε τα κουνούπια, όπως έχει ακουστεί. Υπάρχουν ε, μέτρα ε, υγιεινής που περιορίζουν ε, την εξάπλωση των κουνουπιών. Αλλά εάν αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε εντομοκτώνα δεν θα γνωρίζουμε το τελικό αποτέλεσμα. Θα πρέπει λοιπόν να χρησιμοποιήσουμε σχετικά απλά μέτρα και θα πρέπει να προετοιμαστούμε και εδώ στην Ευρώπη. Έχουμε δει στο παρελθόν ότι μπορεί να υπάρξουν παρόμοιες καταστάσεις και στην Ευρώπη. Για παράδειγμα, όσοι μπουν σε αεροπλάνο για να παρακολουθήσουν τους Ολυμπιακούς Αγώνες θα πρέπει να γνωρίζουν πώς μπορούν να προστατευτούν. Ευχαριστώ κύριε Σπεντιτσίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητοί συνάδελφοι, αναφερόμαστε όλο και περισσότερο στην ανάπτυξη ενός εμβολίου για την καταπολέμηση του ιού του ΖΙΚΑ. Το είπαμε και πριν στην ε, συζήτηση για την ανάπτυξη ενός εμβολίου χρειάζονται αρκετά χρόνια, ενώ για την περίπτωση του ΖΙΚΑ αναφερόμαστε μόνο σε 18 μήνες. Κανονικά αυτό θα έπρεπε να είναι καλό νέο, αλλά 18 μήνες είναι πολύ μεγάλο διάστημα για αποτελεσματική και ταχεία απάντηση στην ε, ε, εκρίζωση του ιού. Ε, το λέω γιατί εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης θα δοθούν περισσότερα κονδύλια για την ε, ανάπτυξη του εμβολίου και στις 8 Φεβρουαρίου ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων σύστησε μια ομάδα εμπειρογνωμόνων για την ε, επιστημονική υποστήριξη ε, ανάπτυξης εμβολίων κατά του ιού Ζήκα τι συνέπειες μπορεί να έχει η εμφάνιση διαφορετικών τύπων του ιού Ζήκα σε ένα καθολικό εμβόλιο. Επίσης, μπορεί να μεταδοθεί από το ένα κουνούπι στο άλλο, από τη μητέρα στο άριο του ε, κουνουπιού. Επομένως, ακόμα και σε αυτή την περίπτωση δεν θα καταφέρουμε να ε, εκριζώσουμε την ασθένεια και δεν θα δώσουμε απλώς περισσότερα χρήματα στις φαρμακοβιομηχανίες και δεν θα εκριζωθεί ο ιός Ζήκα. Επίσης, υπάρχει η τεχνική στήρωση ε, του εντόμου. Ε, μέσω αυτού ε, κυκλοφορεί μεγάλη ποσότητα αρσενικών κουνουπιών που είναι στήρα, που ζευγαρώνουν με άγριες θηλυκές με άγρια φιλικά κουνούπια και στηρώνονται στη συνέχεια και δεν αναπαράγονται. Αυτό αποδείχθηκε ότι ήταν ιδιαίτερο αποτελεσματικό σε άλλη περίπτωση, με άλλα έντομα, το κουνούπι τίγρης στην Αφρική για παράδειγμα. Προσπαθούμε λοιπόν να δούμε κατά πόσον μπορεί να υπάρχουν και άλλοι ή στο δείγμα και ζητάμε γενικότερα να υπάρξει μεγαλύτερη έρευνα στην έρευνα ε, και στη σχέση του ιού Ζήκα ε, με τη μικροκεφαλία ή τη χρήση του υπροξυφένου που θα μπορούσε να είναι και αυτό αιτία της μικροκεφαλίας. Επίσης, ε, ε, θέλουμε να δούμε και έρευνα για την πιθανή μετάδοση του ιού και με άλλες μορφές, για παράδειγμα τη σεξουαλική επαφή ή τη μετάγγιση αίματος. Και επίσης να πω ότι ζητάμε μεγαλύτερη έρευνα ακόμα και στην πρόληψη και στη θεραπεία του ιού, αλλά και κάποιες σημαντικές επιστημονικές αξιολογήσεις για ελαλλακτικές θεραπείες πέραν του εμβολίου, γιατί δεν θα πρέπει για πολλωστή φορά να έχουμε πρόσχημα για να πλουτίσουν οι φαρμακοβιομηχανίες εις βάρος των ασθενών που θα νοσήσουν από τον ιό του Ζήκα. Ο κύριος Παρνιό. Κύριε Πρόεδρε, αγαπητοί συνάδελφοι, καταρχάς θα ήθελα να υπενθυμίσω σε όλους τη διάταξη που θέλαμε να εγκρίνουμε το 2013, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Συμβούλιο, Πρόκειται για την απόφαση που αφορά τις ε, σοβαρές διασυνοριακές απειλές ε, ε, για τους ασθενείς. Ήμουνα εισηγητής και εγκρίναμε τη σχετική διάταξη μετά από αυτά τα οποία διαπιστώσαμε ότι μπορεί να συμβούν με τη γρήπη. των ΙΤΑ 1 εντός εισαγωγικών και το είδαμε και στην Ευρωπαϊκή Επικράτεια και οι διατάξεις όπως έχουν καθοριστεί, υπό τον έλεγχο φυσικά των όσων λέω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ε, μπορούσαν να εφαρμοστούν και για την περίπτωση του έμπολα και νομίζω ότι μπορούν κάλλιστα να εφαρμοστούν και για την περίπτωση του Ζήκα. Πέραν αυτό θα ήθελα επί τη ευκαιρία αυτής της συζήτησης να σας θέσω κάποιες ερωτήσεις, ε, Επιτροπή. Ε, γνωρίζετε ότι πότε η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας ε, θα εκδώσει τη γνωμοδότησή της για τη σχέση μεταξύ ΖΙΤΑ και την ε, συγγενή δυσμορφία ε, του εγκεφάλου των εμβρίων και επίσης ε, ε, τι κονδύλια θα δοθούν και τι έχει δοθεί από αρχές Φεβρουαρίου του τρέχοντος. Αρκούν αυτά τα κονδύλια αν διαπιστωθεί ότι όντως ο ιός οδηγεί ε, και σε νευρολογικές ασθένειες ε, από τους ανθρώπους που μολύνονται, καθώς επίσης και τις προφανείς ενδείξεις που φαίνεται να έχουν σχέση με τον ιό. Επίσης, πώς εξελίσσεται η διαδικασία μετά τη διαπίστωση της ε, νόσου. Τι εξελίξεις έχουμε σε θέματα έρευνας για εμβόλιο, θεραπείας και πότε μπορούμε να ελπίζουμε να ξεκινήσουν αυτές οι κλινικές μελέτες σε μεγάλη κλίμακα. Και τελευταία ερώτηση, στις Φεβρουαρίου ανακοινώσατε ότι θα υπάρξει μια ιατρική ε, μονάδα που θα μπορεί να κινητοποιήσει πόρους. Ε, μπορείτε να μας πείτε για αυτό το νέο ιατρικό σώμα το οποίο θα ε, μπορεί να κινητοποιηθεί για διάφορες επίγουσες ανάγκες. Πότε θα είναι σε εφαρμογή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να κάνω δύο βασικές ε, απλές διαπιστώσεις. Πρώτα απ' όλα, ακούμε συχνά στο δημοσίο διάλογο και στον τύπο το διαβάζουμε ότι ο ιός Σίκα δεν επηρεάζει την Ευρώπη. Από γεωγραφικής απόψεως είναι ορθό υπό την έννοια ότι δεν έχει υπάρξει ακόμα εξάπλωση του ιού στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Ωστόσο, υπάρχουν πληθυσμοί ευρωπαϊκοί στην Γουινέα, στη Γουιάννα, συγγνώμη, στις Γαλλικές Αντίλες, στο Σαμαχτά, σε γαλλικές υπερπόντιες ε, περιοχές δηλαδή, που έχουν ήδη επηρεαστεί. Ευρωπαίοι πολίτες είναι και αυτοί. Επίσης, το 2005-2006 το νησί της ε, Ρεουνιό είχε πληγεί από επιδημία ε, ε, η οποία έχει πλήξει το 40% του πληθυσμού του, δηλαδή μια μαζική επιδημία. Και σήμερα ούτε ένα περιστατικό σε κουνκουνιά δεν έχουμε στο, στη Ρεϊουνιόν. Το οποίο σημαίνει ότι οι αρχές της Γαλλίας σε συνεργασία με τις αρχές της Ρεϊουνιόν εφήρμοσαν μια σειρά βέλτιστων πρακτικών, εφήρμοσαν μια σειρά μέτρων για να αντιμετωπίσουν αυτήν την επιδημία, αυτό το, την ασθένεια που είχε ξεκινήσει να ε, εξαπλώνεται με ραδεύδες ρυθμούς. Και πιστεύω ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μπορεί να αξιοποιήσει το δίκτυο που έχει δημιουργηθεί και ε, υφίσταται σήμερα μεταξύ της ε, Γαλλίας και των υπερπόντιων περιοχών της, να ε, εξετάσει πώς λειτουργεί αυτό το δίκτυο και να το αξιοποιήσει βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να αντιμετωπιστεί η εξάπλωση και η επιδημία του ιού ΣΥΚΑ έτσι ώστε να μην πληγούν οι Ευρωπαίοι πολίτες που βρίσκονται στις υπερπόντιες ε, περιοχές της Γαλλίας. Η κυρία Γκοντίν. Η πολιτική μας ομάδα υποστηρίζει προφανώς το προσχέδιο ψηφίσματος η κίνηση των εμπορευμάτων και των ανθρώπων φυσικά ε, σήμερα ε, ευνοεί την μεγαλύτερη εξάπλωση επιδημιών ε, όπως ο ιός, του, όπως Επίσης, πρέπει να μην ξεχνάσουμε και να μην ξεχνάμε πόσο δραματική είναι η κατάσταση με τη μικροκεφαλία, αλλά επίσης δεν έχει αποδειχθεί ότι έχει προκληθεί από τον ιό, του, από Ένα ποσοστό ε, των ε, γυναικών που έχουν γεννήσει παιδιά με μικροκεφαλαία ήταν φορείς του Ιούζικα. Μπορεί να οφείλεται σε άλλα αίτια. Ε, κάποιου συνδρόμου ή γενετικά. Στην Κολομβία υπήρξε μια έξαρση ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείε έχουμε παράλληλη έξαρση μάλλον στην Κολομβία του Ιουσίκα και ε, γεννήσεων με μικροκεφαλία, ενώ στις Ηνωμένε Πολιτείε χωρίς να υπάρχουν περιστατικά ε, του Ιουσίκα είχαμε 25 ε, περιστατικά το χρόνο μικροκεφαλίας. Επομένως θα πρέπει να γίνει μεγαλύτερη και εις βάθος έρευνα επιστημονική για το κατά πόσον τελικά συνδέεται ο ιουσίκα με τη μικροκεφαλία ή φταίει κάτι άλλο. Οι βραζιλιάνικες αρχές έχουν ε, επιβάλει την χρήση της προφύλαξης ε, και με αυτόν τον τρόπο απαγόρευσαν την, ε, του και προτίθεμε να υποβάλω σχετική τροπολογία στο ψήφισμα με το οποίο θα ζητήσετε την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κάνει το ίδιο. Και πάλι για στην Ευρώπη με βάση την αρχή της προφύλαξης. <clears throat> Κύριε δεν έχω να προσθέσω πολλά σε αυτά που είπαν οι συνάδελφοι. Πρέπει να κάνουμε ό,τι περνάει από το χέρι μας για να σταματήσει η εξάπλωση του ιού. Η Βραζιλία είναι μια από τις χώρες που έχουν πληγεί περισσότερο και γνωρίζουμε ότι στη Βραζιλία θα γίνουν οι Ολυμπιακοί Αγώνες το καλοκαίρι που μας έρχεται. Επομένως γνωρίζουμε ότι ε, χιλιάδες άνθρωποι θα πάνε στην Βραζιλία, θα επισκεφτούν τη Βραζιλία για τους αγώνες. Που σημαίνει ότι ο κίνδυνος εξάπλωσης του ιού με αυτές τις μετακινήσεις είναι τεράστιος. Προς τις Ηνωμένε Πολιτείες, οι οποίες πρόσφατα μάλιστα ανακοίνωσαν ότι οι αθλητές τους έχουν το δικαίωμα να αποφασίσουν ε, μόνοι τους και εάν θεωρήσουν ότι ο κίνδυνος είναι υπερβολικά υψηλός, ε, έχουν το δικαίωμα οι αθλητές των ΗΠΑ να μην συμμετάσχουν στους Ολυμπιακούς Αγώνες. Το ότι θα διεξαχθούν λοιπόν οι Ολυμπιακοί Αγώνες στη Βραζιλία ε, κάνει τα πράγματα ακόμα πιο επικίνδυνα, το οποίο σημαίνει ότι πρέπει όσο το δυνατόν γρηγορότερα και εμείς να λάβουμε τα μέτρα μας. Ο πρώτος, ευχαριστώ. Και τώρα θα δώσουμε το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή για να απαντήσει σε όλες αυτές τις παρατηρήσεις των Ευρωβουλευτών. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα να κάνω κάποιες παρατηρήσεις σε σχέση με το ψήφισμα. Καταρχάς το διεθνές πλαίσιο για τις διασυνοριακές απειλές ε, είναι η Διεθνής Σύμβαση του ΠΟΗ. Την 1η Φεβρουαρίου φέτος ο ΠΟΗ λόγω της εμφάνισης του ιού ε, κήρυξε κατάσταση έκτακτης ανάγκης και κινητοποιήθηκαν οι ε, σχετικοί μηχανισμοί για να αντιμετωπιστεί η εμφάνιση της επιδημίας. Ο κύριος Παρνιό είπε ότι σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης από το 2013 έχουμε απόφαση Συμβουλίου και Κοινοβουλίου για τις διασυνοριακές απειλές υγείας. για την αντιμετώπιση τέτοιων απειλών σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και αυτός ο μηχανισμός κινητοποιήθηκε ε, Συγκλήθηκε δηλαδή η ε, Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας ε, που έχει συζητήσει επανειλημμένα το θέμα και έχουμε ζητήσει από το ΕΚΠΕΝ να εκπονήσει μελέτη αξιολόγηση κινδύνου Αυτές οι αξιολογήσεις ε, κινδύνου εξετάζουν τις συμβουλές προς το κοινό, τις ε, συμβουλές προς τους ε, επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, την, το σενάριο που θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί, την εξέταση προβλημάτων δυσμορφιών κλπ και καθώς ε, και θέματα που συνδέονται με τις ε, μεταφορές ε, και με τον περιορισμό των φορέων. Ήδη είχαμε εις βάθος συζήτηση πάνω στο σχέδιο κειμένου του ΕΚΠΕΝ και θα πραγματοποιηθεί άλλη συνάντηση της Επιτροπής αύριο για να συζητήσουμε τη δημοσίευση του κειμένου εντός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Υπάρχει σύγχυση όσον αφορά ιδιαίτερα τις ε, συμβουλές προς ε, ταξιδιώτες. Θα δημοσιευτούν δηλαδή συγκεκριμένες οδηγίες. Επίσης, Έχουμε κινητοποιήσει ένα δίκτυο που έχουμε στο ε, Κοινό Κέντρο Ερευνών σχετικά με ε, τις ε, συγγενείς λοιμώξεις για να εξεταστούν οι δυσμορφίες που συνδέονται με την εξάπλωση του ιού Και μπορώ επίσης να σας πω ότι έχουν ληφθεί μέτρα στο πλαίσιο της ευρωπαϊκής νομοθεσίας για ε, για τους ε, ε, αιματοδότες και για τις χορηγίες οργάνων. Και επίσης, η Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας ζήτησε από το ΕΚΠΕΝ να εκπονήσει ερωτηματολόγιο προς τα κράτη-μέλη. Η δουλειά αυτή συνεχίζεται αυτή τη στιγμή. Ε, οι πληροφορίες μου λένε ότι υπάρχουν 72 εργαστήρια σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης που έχουν την δυνατότητα να εντοπίζουν τον ιό Ζήκα σε 23 κράτη-μέλη. Θα πρέπει να δούμε πώς μπορεί να ε, γίνει μοίρασμα των υποδομών ώστε να καλυφθούν και τα υπόλοιπα κράτη-μέλη. Όσον αφορά την ανάπτυξη εμβολίων και θεραπείων, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός ε, Φαρμάκων στις 8 ε, Φεβρουαρίου δημιούργησε μια ειδική ομάδα ε, για την παροχή συμβουλών σχετικά με τον ιό Ζήκα. Κατόπιν έχουμε το θέμα του ελέγχου των φορέων. Είχαμε πείρα στο θέμα αυτό σε σχέση με άλλους ιούς εντός της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης. Διάφορα κράτη-μέλη, όπως υπόθηκε, έχουν πείρα στο, ε, στον τομέα αυτό, ιδιαίτερα η Ελλάδα, η Ιταλία και η Γαλλία. Ε, και η ίδια η Γαλλία και, η, και τα υπερπόντια εδάφη, όπως άλλωστε και η Ισπανία και η Πορτογαλία. Θα μπορούσα επίσης να αναφέρω ότι το ΕΚΠΕΝ και έχουμε εδώ την Διευθύντρια έχει δημιουργήσει δίκτυο για τις ε, ασθένειες που μεταδίδονται μέσω φορέων και θέλει να δημιουργήσει σχετικό ευρωπαϊκό δίκτυο. Τέλος, Όσον αφορά την απειλή από τα κουνούπια, μπορώ να αναφέρω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση είναι σημαντικός χορηγός του Διεθνούς Ταμείου ε, που έχει ε, προμηθεύσει πολλές ε, κουνουπιέρες για την προστασία ανθρώπων από τους ιούς που μεταφέρουν τα κουνούπια. Όσον αφορά την κινητοποίηση ειδικών γιατρών από την Ευρωπαϊκή Ένωση, δεν υπήρξε έτοιμα μέχρι στιγμής. Υπάρχει όμως ο μηχανισμός. Υπάρχει το προσωπικό. Εάν υπάρξει ανάγκη λοιπόν, θα μπορέσουν να συμβάλλουν. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι πρόκειται για μια κατάσταση εν εξελίξη. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όμως ήδη έχει θεσπίσει εντός του, παρόντος, του νομοθετικού πλαισίου μέτρα για να αντιμετωπιστεί η κρίση αυτή. Ευχαριστώ. Εγώ σας ευχαριστώ. Πριν ε, δώσω το λόγο στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και στο Κέντρο Πρόληψης Νόσων, αν θέλουν να προσθέσουν κάτι, υπάρχει μια επιπλέον ερώτηση από την κυρία Ριβαζή. Ναι, ευχαριστώ για τις απαντήσεις σας. Κάπου νομίζω δεν απαντήσατε σωστά σε όλα τα σημεία. Ε, επειδή ο Ζήκα είναι πραγματικά διεθνής ε, απειλή για την υγεία, ε, διότι στο Νότια Ευρώπη έχουμε Ισπανία, Ιταλία, Γαλλία που θα έχουν κουνούπια το καλοκαίρι και θα βρεθούμε αντιμέτωποι με τέτοια προβλήματα. Είπατε ότι δεν υπάρχει εμβόλιο, αλλά ε, μόλις έμαθα ότι υπάρχει ένα ειδικό εργαστήριο, το Bara Biotech, το οποίο ανέπτυξε δύο εμβόλια, τα οποία πρέπει ακόμα να ε, ελεγχθούν για την αποτελεσματικότητά τους ως προς την ασφάλεια. Τι συμβαίνει με αυτό το ε, ειδικό εργαστήριο. Δεύτερον, μας λέτε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ε, κινητοποίησε 10 εκατομμύρια ευρώ, ενώ ε, εγώ από ό,τι γνωρίζω ζήτησαν κονδύλια κάποιοι Αργεντίνοι ερευνητές ε, ε, δεν ξέρω κατά πόσον οφείλεται σε κάποιο κοκτέιλ ή σε κάτι άλλο για με το περι, για την μικροκεφαλία. Και επίσης υπάρχουν κάποια ερωτηματικά για ένα εμβόλιο ε, για διφθερίτιδα και τέτανο που δόθηκε σε πολλές ε, γυναίκες από τη Βραζιλία. Δεν έχω φυσικά απαντήσει σε όλα αυτά, αλλά θα ήταν ενδιαφέρον να γίνουν κάποιες μελέτες επ' αυτού για να ε, αποκλείσουμε αυτές τις παραμέτρους. Υπάρχει πολύ μεγάλο ενδεχόμενο να οφείλεται στο ζήκα η μικροκεφαλία και κάτι τελευταίο στις συστάσεις. Κανείς δεν ε, αναφέρεται στα μέσα τα οποία υπάρχουν για την παρακολούθηση των εγγύων. Γιατί σε αυτές τις χώρες ε, πολύ ωραία και καλά να λέμε μη πάτε, αλλά υπάρχουν επιτόπου πολλές έγκυες γυναίκες. Παρακολουθούνται τι γίνεται με τις εκτρώσεις, γιατί ε, απαγορεύεται η άμβλωση ε, στη Βραζιλία. Τι γίνεται λοιπόν όταν οι γυναίκες αυτές έχουν έμβρια με μικροκεφαλία. Πρέπει ε, να δούμε αν επιτρέπεται η άμβλωση σε αυτή την περίπτωση και επίσης τι εξελίξεις υπάρχουν όσον αφορά την αντισέλιψη και τα κέντρα αναπηρίας. Διότι από ό,τι φαίνεται ο ιός απέδειξε ότι υπάρχει ένα ε, θέμα ε, διανοητικής ανάπτυξης και θα έχουμε λοιπόν πολύ περισσότερους αναπήρους ε, και για την ε, μικρο... Ε, πέραν από τις μικροκεφαλίες. Τι γίνεται λοιπόν με τις εγγύους πέραν από τις, ε, τους ανθρώπους που, στους οποίους συμβουλεύουμε να μην πάμε. Μην ξαναρχίσουμε ερωτήσεις. Κύριε Φαρία, έχετε δει το λόγο, αλλά σύντομα. Ναι κύριε Πρόεδρε, πολύ σύντομα. Συνεχίζω από αυτά που λέει η κυρία Ριβαζή. Δεν συζητήθηκαν εδώ όλα τα θέματα. Ε, το περιπροξηφέν είναι ένα από τα θέματα τα οποία ζήτησαν να συμπεριληφθούν στο ψήφισμα ε, και κατάφερα να αναφερθεί παρά το γεγονός ότι διαφωνούσαν κάποιες πολιτικές ομάδες. Ε, υπάρχουν κάποιες περιπτώσεις στη Βραζιλία που αποδείχθηκε ότι ε, κατά πάσα πιθανότητα η μικροκεφαλαία προέρχεται από το ε, βίρους, από τον ιό Ζήκα και Υπάρχει και ένα εντομοκτόνο το οποίο αποφασίστηκε από το δήμαρχο μιας περιοχής να χρησιμοποιηθεί στο πόσιμο νερό, γιατί χάρη στο πόσιμο νερό ε, μολύνονται, μάλλον όχι χάρη εξαιτία του πόσιμου νερού μολύνονται οι αγίες γυναίκες. Ευχαριστώ. Να δώσουμε και πάλι το λόγο στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και μετά στην Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και στο Κέντρο Πρόληψης Νόσων. Ευχαριστώ για την ερώτηση. Όσον αφορά τη σχέση με τα εμβόλια τα οποία ε, χορηγούνται στα παιδιά και τις γενετικές αυτές ανομαλίες, ε, δεν ε, υπάρχουν εκθέσεις που σχετίζουν τα εμβόλια των παιδιών ε, με τέτοια προβλήματα. Αν υπάρχουν τέτοιες πληροφορίες ε, επ' αυτού θα τα εξετάσουμε μαζί με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων και το αυτό ισχύει και για τα ειδικά εμβόλια τα οποία αναφέρθηκαν. Αν όντω ε, υπάρχουν πληροφορίε που σχετίζονται με εμβόλια ή πιθανέ θεραπείε, αυτό σίγουρα μα ενδιαφέρει και θα το παρακολουθήσουμε. Όσον αφορά τις ε, εικασίες στον τύπο για το εντομοκτόνο αυτό το οποίο αναφέρθηκε και σχετίζεται με τη μικροκεφαλία, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν έχει αποδείξεις που να υποστηρίζουν τις απόψεις που εκφράζονται στα άρθρα αυτά το εντομοκτώμα αυτό ε, δεν γνωρίζουμε να δημιουργεί γενετικές ανομαλίες, δεν υπάρχουν αρκετές επιστημονικές ενδείξεις ε, που ε, να υποστηρίζουν αυτή την άποψη ότι υπάρχει σχέση με τη χρήση των εντομοκτώνων και αυτών των γενετικών ανομαλιών. Όσον αφορά τα κονδύλια τα οποία διατίθενται για την έρευνα, ανέφερα το ποσό αυτό των 10 εκατομμυρίων, αλλά σας είπα επίσης ότι Υπάρχουν ναι, προγράμματα εξελίξη τα οποία κατά πάσα πιθανότητα θα μπορέσουν να χρησιμοποιηθούν και να υπάρξει ένα ποσό 65 εκατομμυρίων ευρώ σε διάφορες περιοχές σε σχέση με το δάγκιο πυρετό ε, και μέτρα για επιτήρηση και έρευνα. Τα 10 λοιπόν αυτά εκατομμύρια δίνονται επιπλέον των 65 ε, περίπου εκατομμυρίων που διατίθενται για άλλα ερευνητικά προγράμματα τα οποία έχουν σχέση με την επιδημία. Όσον αφορά την ερώτηση της κυρίας ε, Ριβαζή για την ε, φροντίδα των εγγύων γυναικών στην Νότια Αμερική, αυτό είναι σαφώς ευθύνη της, ε, των χωρών της Νότιας Αμερικής ε, και φυσικά σε συνεργασία με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας. Η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας έχει εκδώσει κατευθυντήριες γραμμές, έχει δώσει και κάποιες συμβουλές οι οποίες σε γενικές γραμμές συνάδουν με τα όσα υποστηρίξαμε και εμείς ε, στην αρμόδια επιτροπή μας και επομένως είναι ευθύνη της κάθε χώρας στην Νότια Αμερική κατά πόσον θα λάβουν υπόψη αυτές τις συμβουλές και θα τις εφαρμόσουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. κύριος Μπερτολίνη. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Και εγώ θα ήθελα να κάνω ορισμένες παρατηρήσεις για κάποια από τα πράγματα που υπόθηκαν από ευρωβουλευτές σε σχέση με την Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και επίσης πώς και πότε έγινε η συσχέτιση μεταξύ του ιού Ζήκα ε, και της μικροκεφαλίας. Αυτό είναι κάτι το οποίο ακόμα εξετάζεται. Εγώ θα ήθελα πρώτα απ' όλα να αναφερθώ στη δήλωση του κ. Ε, Bruce Όλουικ, ο οποίος είναι υπεύθυνο ε, στον ΠΟΗ ε, για τον έλεγχο της επιδημίας του ΖΙΚΑ, ότι στον τομέα της υγείας όλοι είναι ένοχοι μέχρι να αποδείξουν την αθωότητα τους. Είναι δεύτερη φορά που διαπιστώνεται μια επιδημία μικροκεφαλίας σε συνδυασμό με τον ιό Ζήκα. Έχει ξαναυπάρξει ε, τέτοιο, τέτοια περίπτωση στη Γαλλική Πολυνησία με 18 περιστατικά, αν θυμάμαι καλά. Έχουμε 280 ε, περιστατικά όπου διαπιστώθηκε ε, ότι, ο φορέας του ιού, ε, ότι η φορέας του ιού γέννησε παιδί με μικροκεφαλία και πρέπει να το συγκρίνουμε αυτό τον αριθμό με τα 163, 163 ε, ε, περιστατικά μικροκεφαλία στον χρόνο. Επίσης, έχουν παρατηρηθεί ε, έχει παρατηρηθεί, έχει εντοπιστεί μάλλον η ΩΣΥΚΑ στην Σλοβενία και σε μία-δύο άλλες χώρες ε, στο ε, αμνιακό υγρό εγγύων. Πιστεύω ότι ο λόγος που δεν, έχει, δεν έχουμε ακόμα άλλα περιστατικά είναι ότι η μικροκεφαλία διαπιστώνεται, διαγνώσκεται αργά συνήθως σε προχωρημένο στάδιο της εγκυμοσύνης πολλές φορές ακόμα και ε, κατά τη γέννα. Το οποίο σημαίνει ότι αν η επιδημία έχει ξεκινήσει το 2015 του ιού του ΣΥΚΑ είναι λογικό να μην έχουμε ακόμα ε, πολλά περιστατικά μικροκεφαλίας που να οφείλονται σε ιό να μην έχουν διαγνωστεί. Ο επιπολασμός της μικροκεφαλίας είναι 2,5 ε, περιστατικά ανά 10.000 ε, νεογνά στην Ευρώπη. Το οποίο σημαίνει ότι είναι πάρα πολύ σπάνιο. Ε, αυτό συμπεριλαμβάνει και τις, τις αμπλώσεις. Και πρέπει να το λάβουμε υπόψη μας. Όσον αφορά τώρα την σύνδεση για, με το εντομοκτόνο πυροπροξυφέν, εχθές οι πόοι ε, και με τον εμβολιασμό μάλλον, εξέδωσε χτε μια δήλωση. Πρώτα απ' όλα, όσον αφορά τον παιδικό εμβολιασμό, δεν υπάρχει κάποια επιστημονική απόδειξη ότι το εμβόλιο αυτό το οποίο χρησιμοποιείται επί δεκαετίε σε ολόκληρο τον κόσμο προκαλεί μικροκεφαλία. Αυτό για, το για τον εμβολιασμό, για το εμβόλιο. Κάτι αντίστοιχο θα μπορούσε κανεί να πει για το ε, το οποίο προσυδειάζει σε μία ουσία, μία ορμόνη που ε, υπάρχει μόνο στα σπονδυλωτά και στα σπόνδυλα και δεν έχουμε ε, κανένα επιστημονικό δεδομένο το, οποίο να συντείνει στο ότι το η πύρη προξηφέν προκαλεί τερατογενέσεις ή γενετικές ε, μεταλλάξεις. Ε, είναι... Γνωρίζουμε ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε εργαλεία στη διάθεσή μας για να καταπολεμήσουμε την εξάπλωση του ιού του, ε, των φυσικών φορέων του τοκουνουπιών και έχουμε ξεκινήσει να κατηγορούμε τις διάφορες ε, ε, ανά τον κόσμο. κάποιε κυβερνήσει έχουν ξεκινήσει να το κάνουν, αλλά εγώ θέλω να επισημάνω και να, να επιστήσω την προσοχή σα ότι πρόκειται για μετα, ε, ε, ασθένειες οι οποίες μεταδίδονται μέσω ξενιστών. Και εκεί εστιάζουμε τις προσπάθειές μας, προσπάθειες περιορισμού της ξάπλωσης των ξενιστών του ιού. Τώρα, Βεβαίω χρειάζεται περισσότερη έρευνα και για τα διαγνωστικά εργαλεία, το είπαν και οι πολλοί ομιλητέ, για την πιθανότητα να δημιουργηθεί κάποιο εμβόλιο κατά του Ιουζίκα. Εδώ θέλω να διευκρινίσω το εξή για τα εμβόλια. Ο ΠΟΗ έχει εκτιμήσει ότι θα χρειαστούν 18 μήνες για την πρώτη πειραματική φάση ενός πιθανού εμβολίου. Δεν μιλάμε για 18 μήνες μέχρι τη στιγμή που θα είναι διαθέσιμο για να χρησιμοποιηθεί σε ανθρώπους ε, και να ε, παραχθεί εμπορικά. Ε, Επίση, όσον αφορά τη χρηματοδότηση, η ΠΟΕ, η έχει ζητήσει 56 εκατομμύρια δολάρια για τους επόμενους 6 μήνες, 25 για τον ΠΟΗ και την Παναμερικανική Οργάνωση Υγείας και τα υπόλοιπα για άλλες οργανώσεις υγείας ε, για να γίνουν καμπάνιες ευαισθητοποίησης ε, ανά τον κόσμο στις περιοχές που πλήττονται. Η ευαισθητοποίηση είναι πάρα πολύ σημαντική ακόμα και αν αυτό δώσει τη δυνατότητα, ακόμα και αν μια κυβέρνηση μάλλον καταφέρει ε, να απολυμάνει μια ολόκληρη περιοχή, ένα κουνούπι το οποίο επιβάζεται και επιβιώνει σε μια λιμνούλα, στο μπαλκόνι σας, σε ένα ποτήρι, μπορεί να δημιουργήσει προβλήμα, μπορεί να, εξαπλω... να συντείνει στην εξάπλωση του ιού. Αυτά από πλευράς μας κύριε Πρόεδρε, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Το ΕΚΠΕΝ. Θα ήθελα να επανέλθω σε κάποια από τα θέματα αυτά. Καταρχάς αναφέρθηκε ότι Υπάρχει εμπειρογνωμοσύνη στην Ευρώπη για την αντιμετώπιση των νόσων που μεταφέρουν τα κουνούπια. Αυτό είναι αλήθεια. Ανέφερα σήμερα το πρωί ότι οι χώρες όπου υπάρχουν ε, αυτοί οι φορείς των νόσων έχουν επιρογνωμοσύνη για την ε, αντιμετώπιση διαφόρων από αυτές τις νόσους και θα χρησιμοποιήσουμε αυτή την επιρογνωμοσύνη. Για παράδειγμα, όπως είπε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας, ε, μπορούν όλες οι χώρες αυτές να ανταλλάσσουν εμπειρογνωμοσύνη και εμπειρίες. Έχουμε δίκτυο εντομολόγων που μελετούν τα κουνούπια αυτά. Και όπως είπα σήμερα το πρωί, θα πρέπει τώρα να παρακολουθήσουμε την κατάσταση όσον αφορά την παρουσία των ιών στην Ευρώπη και να ελέγχουμε και όσους εισέρχονται στην Ευρώπη, ιδιαίτερα όταν προέρχονται από περιοχές όπου υπάρχουν τα κουνούπια αυτά. Αυτό θα συζητήσουμε αύριο στην Επιτροπή Υγειονομικής Ασφάλειας. Όσον αφορά τον ιό του Δυτικού Νείλου, χαρτογραφήσαμε την κατάσταση, επικαιροποιούσαμε τους χάρτες, ώστε να είναι πάντα διαθέσιμες οι πληροφορίες σχετικά με το που υπάρχει κίνδυνος. Πού βρίσκονται οι φορείς ε, της νόσου και ποιες είναι οι επικίνδυνες περιοχές της Ευρώπης. Θα ήθελα να επανέλθω στο θέμα της έρευνας. Φυσικά πρέπει να συλλέξουμε περισσότερα στοιχεία σχετικά με τον τρόπο μετάδοσης. Αυτό που χρειαζόμαστε τώρα όμως είναι πληροφορίες για να ποσοτικοποιήσουμε τον κίνδυνο. Ξέρουμε ότι υπάρχει κίνδυνος ε, για τις εγγύους το παιδί να γεννηθεί με μικροκεφαλία, αλλά δεν ξέρουμε πόσο μεγάλο είναι αυτός ο κίνδυνος. Αυτό ισχύει για κάθε έγκυο γυναίκα, για το 10% για το 30% των ε, περιπτώσεων. Τέτοιε μελέτε εκπονούνται αυτή τη στιγμή ώστε να μπορέσουμε να ποσοτικοποιήσουμε τον ε, κίνδυνο. Το ίδιο ισχύει με τη σεξουαλική μετάδοση. Έχουμε δύο τεκμηριωμένες περιπτώσεις. Δεν ξέρουμε όμως πόσο συχνά ε, γίνεται η σεξουαλική μετάδοση. Και τέλος θα ήθελα να αναφερθώ στην Ρεϊνιόν. Το 40% του πληθυσμού το 2005 με 2006 είχε ε, ε, ε, μολυνθεί από τον ιό. Αλλά δεν υπήρχε ανοσία Και αυτό ακριβώς ε, αντιμετωπίζει και η Βραζιλία αυτή τη στιγμή, ότι κανείς δεν έχει έρθει σε επαφή με τον ιό, άρα δεν ε, έχει αναπτύξει κανείς ανοσία. Ε, αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει πια ο ιός τσικουγκούνια στην Ρεϊνιό και αυτό έχει να κάνει και με το γεγονός ότι έχει αναπτύξει ανοσία πολλοί κόσμος. σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε εργαστήρια ικανά να διαγνώσουν τον ιό. Τα κράτη-μέλη που δεν έχουν τέτοια εργαστήρια έχουν συμφωνίες με γειτονικέ χώρες για την πραγματοποίηση διαγνώσεων. Πιστεύουμε λοιπόν ότι υπάρχει επαρκές δυναμικό στην Ευρώπη για την διάγνωση των λοιμόξεων αυτών. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ για τις παρατηρήσεις σας και τις απαντήσεις σας. Κυρία Φαρία, θέλετε και πάλι το λόγο. 30 δευτερόλεπτα. Για τον κύριο Μπερτολίνη, δεν ήξερα ότι ήσασταν εδώ, αλλά κύριε Μπερτολίνη, το πυροπρόξιφάι δεν επιτρέπει στο κουνούπι να μεγαλώσει, να γίνει ενήλικο και να αναπαραγεί και να μεταφέρει ασθένειες. Η μικροκεφαλία σημαίνει μικρός εγκέφαλος. Δεν ξέρω, δεν είμαι επιστήμονας. Απλώς θα ήθελα να ξέρω ε, πώς μπορούμε να προστατεύσουμε τη δημόσια υγεία. Είπατε ότι αντίθετα με την αρχή που ισχύει στο δίκαιο, στο Ιντούμπριο Προρέο, ε, δεν θα πρέπει να θεωρείτε ότι ο πυροπροξυφένη είναι ένοχο ε, μέχρι να αποδειχθεί η αθότητα του, ο κύριος Μπερτολίνη. Δεν είπα κάτι τέτοιο. Απλώς ανέφερα μία φράση του γενικού μας διευθυντή, ο οποίος εξετάζει τα θέματα αυτά, ο οποίος είπε ότι η σχέση μεταξύ του ιού Ζήκα και της μικροκεφαλίας θα πρέπει να θεωρείται πραγματική μέχρι να αποδειχθεί ότι δεν υπάρχει σχέση. Αλλά αυτό αποτελεί απλώ πρόκληση για να πούμε ότι έχουμε σοβαρές ενδείξεις να πιστεύουμε ότι ο ιός Ζήκα προκαλεί μικροκεφαλία σε αυτή την περίπτωση. Επομένως ε, εδώ ε, έγινε το θέμα, αυτό πιστεύει η Παγκόσμια Οργάνωση Υγείας και αυτή είναι η επίσημη θέση της οργάνωσης. Ωραία, θα ολοκληρώσουμε τη συζήτησή μας. Ε, κάποιες τελευταίες πληροφορίες για τη συζήτηση αυτή. Η ημερομηνία κατάθεσης τροπολογιών 25 Φεβρουαρίου, 12 το μεσημέρι, μόνο στα αγγλικά. Αυτά λοιπόν είχα να σας πω. Και με αυτό ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη. Εμείς βέβαια δεν έχουμε εξαντληθεί, μόνο η μερίσια διάταξη εξαντλήθηκε. Θα μπορούσαμε να συζητήσουμε ε, και να περάσουμε σε άλλες δραστηριότητες. Ευχαριστώ για την προσοχή σας και τη συμμετοχή σας.